Good afternoon, colleagues. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Α ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μα. Ξεκινάμε με την έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Σα ευχαριστώ. Περνάμε ευθύ αμέσω στο σημείο 3 τη ημερήσια διάταξη, καθότι δεν έχω ανακοινώσει να κάνω να καλωσορίσω τους συμμετέχοντες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον κύριο Κεραμουσού και τον κύριο Ουρέλ από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού και τον κύριο Χίντον και τον κύριο Κεριόν Κασόνη, καθώς επίσης και την κυρία Μάτσεν από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ. Η συνεδρία αυτή μεταδίδεται μέσω διαδικτύου και διοργανώνεται από κοινού από τις ε, δύο καθήλυνα αρμόδιες επιτροπές στα πλαίσια του κανόνα του άρθρου 55 μάλλον του κανονισμού που προβλέπει κοινέ ε, συνεδριάσεις των δύο αυτών επιτροπών για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Βασιζόμαστε στην, στο άρθρο 54 λοιπόν του κανονισμού συμμετέχουν επίσης η Ίτρε και η Τραν και η Ρέτζι Έκον Αύκο Όλες αυτές οι κοινοβουλευτικέ επιτροπές καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτή τη συνεδρίαση. Έχει καθαρά τεχνική φύση η συνεδρίαση αυτή. στόχος μας είναι να προσαφηνίσουμε ορισμένα στοιχεία του σχεδίου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λάβαμε χθε απαντήσεις τις 110 ερωτήσεις που είχαν υποβάλει οι Ευρωβουλευτές. Πρόκειται προφανώς για απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στείλαμε εμεί ερωτήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απάντησε σε ερωτήσεις αυτές ότι είχε λιγότερο από μία εβδομάδα. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να θέσουν ε, ή δυνατόν νέα ερωτήματα σε σχέση με τις γραπτές αυτές ερωτήσεις που έχουμε στο έγγραφο. Εκτός βέβαια και αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις που σας έχουν δοθεί για να απαιτείτε περαιτέρω διευκρινήσεις. Ας δώσω τώρα στον Συμπρόεδρο την, το λόγο για να εξηγήσει το πώς θα λειτουργήσουμε. Ευχαριστώ Ροπέρτο. Να συμπληρώσω ίσως ε, για τις ειδικέ ερωτήσεις από την Επιτροπή Μεταφορών και Βιομηχανίας. Έχουμε προσώπους υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις Γενικές Διευθύνσεις MOVE και Research ε, μεταφορών και έρευνας. Η διαδικασία είναι όπως ε, την περιέγραψε ο Ρομπέρτο. Ουσιαστικά σήμερα πρόκειται κατά κύριο λόγο για μια τεχνική συνεδρίαση ε, μέχρι να φτάσουμε στην κανονική διαδικασία. Δηλαδή, σε ερωτήσεις παρακαλείστε να μην κάνετε πολιτικές δηλώσεις, ούτε δύο, πάνω από δύο λεπτά, και να έχει τρία λεπτά στη συνέχεια η Κομισιόν για να απαντά. Και μετά από δύο λεπτά θα σας στέλνω ένα μικρό ακουστικό μήνυμα, βλέπε σφυράκι. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να τηρείτε το χρόνο σας για να μπορέσουν να ρωτήσουν όλοι όσοι το επιθυμούν. Πινκ-πονγκ δηλαδή θα είναι. Όχι μόνο μεταξύ ημών των βουλευτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ λεπτή κατανομή του χρόνου μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οι συγητές παρακαλούνται στην αρχή να μιλήσουν και ως Φερνάντες από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Θέλει να κάνει τελευταία ερώτηση. από την Επιτροπή Προπολογισμού, συγγνώμη, και θα αρχίσει ο κύριος Μπούλμαν από την Οικονομική. Οπότε θα πηγαίνουν ερωτήσει σε ένα λάξ. Έκον μπάτζ, έκον μπάτζ και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντά. Πάντα για θέματα τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και τη Επιτροπή Προπολογισμού. Αν συμφωνείτε, αρχίζουμε λοιπόν και ακούμε πρώτα τον Ούντο Μπούλμαν, εισηγητή τη Επιτροπή ε, Οικονομικών και νοσηματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρό μας και τους συναδέλφους που ήρθατε από τις επιτροπές σας για να παρευρεθείτε στην συζήτηση. Είναι τεχνική ε, είναι για να κάνουμε μια καταγραφή ε, της κατάστασης και να αποκομίσουμε δεδομένα. Εγώ έχω μια ερώτηση που έχει να κάνει με την πρακτική ζωή. Πολλοί ενδιαφέρονται για το τι ε, θα σημάνει στην πράξη αυτό το σχέδιο Juncker. Εμείς έχουμε ως πρόθεση βασική να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική. Παράδειγμα, ευρυζωνικότητα το γρήγορο ίντερνετ, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα για όλη την Ευρώπη. Η ευρυζωνικότητα χωλαίνει σε πολλές χώρες. Για ποιο λόγο, διότι δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και γιατί δεν αποδίδει άμεσα και στις χώρες που λειτουργεί καλά, Γαλλία έδωσε το καλό παράδειγμα, χρειάζονται ιδιωτικά κεφάλαια, χρειάζονται κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και επιπλέον χρήματα από το δημόσιο. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μου πούν τι κάνει μια χώρα σαν την Πορτογαλία που είναι ο συνεισηγητής μου. Πώς θα αναπτυχθεί εκεί η ευρυζωνικότητα στην Ήπεθρο μέχρι και τις περιφέρειες της Πορτογαλίας με τη βοήθεια του νέου μηχανισμού αυτού για το Ταμείο. Πώς θα λειτουργήσει αυτό, ποιος θα πληρώσει ποια ποσά. Με αυτό το παράδειγμα μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλείται να απαντήσει. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να σας εξηγήσουμε σήμερα τις, ε, την πρόταση αυτή. Προσμένουμε να συνεργαστούμε μαζί σας κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ε, και της παρακολούθησης του Ταμείου. Σε ό,τι αφορά την ε, ερώτηση αυτή για τις, τα πρακτικά ζητήματα διαφορών σχεδίων και ιδιαίτερα της ευρυζωνικότητας. Όπως γνωρίζετε, ο κεντρικός πυλώνας της ε, ε, πρότασης είναι η βιωσιμότητα, η οικονομική βιωσιμότητα των σχεδίων. Εμείς θέλουμε να εστιαστούμε σε project τα οποία θα είναι βιώσιμα αλλά θα έχουν μεγαλύτερο του συνήθους κίνδυνο. Ε, το, η ευρυζωνικότητα είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει άμεση κερδοφορία. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ καλός ε, ε υποψήφιος Ε, υπάρχουν ε, και άλλα τέτοια σχέδια τα οποία δίνουν κερδοφορία ε, μακροπρόθεσμα και οι επενδυτές διστάζουν να αναλάβουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα αναλάβει τέτοιου τύπου σχέδια τα οποία είναι μακροπρόθεσμα οικονομικά βιώσιμα έτσι ώστε οι επενδυτές να διευκολυνθούν να επενδύσουν σε σχέδια τα οποία κανονικά δεν θα χρηματοδοτούνται από τις αγορές. Εγώ άλλο ρώτησα, αν μπορώ να επιμείνω. Ε, στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό, ποιος θα μπορούσε να συγχρηματοδοτεί, ποιος θα ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ο ρόλος των ιδιωτών επενδυτών και των δημοσίων ε, επενδύσεων, από το δημόσιο κορβανά, αυτό ρώτησα. Ε, το επέτρεψε αυτό, λέει ο πρόεδρος, γιατί δεν είχε εξαντλήσει το δίλεπτο ο Μπούλμαν. Κατά τα άλλα, ε, ας προσπαθήσουμε να μην έχουμε τέτοιες συνομιλίες, γιατί θα υπάρξουν προβλήματα και δυσκολίες χρονικές. Ευχαριστώ. Από πρακτικής ε, πλευράς, οι προτείνοντες θα πάνε στο ταμείο και θα προταθεί η καταμερισμός της χρηματοδότησης μεταξύ του Ταμείου Ιδιωτών και ενδεχομένως και κρατικού τομέα. Το Ταμείο ε, θα προσπαθήσει να είναι καταλή ιδιωτικές επενδύσεις, οπότε ε, θα αναλάβει το, υψηλότερο, το κομμάτι που αντιστοιχεί στον υψηλότερο κίνδυνο της επένδυσης. Το κομμάτι που αντιστοιχεί στον υψηλότερο κίνδυνο, το πιο επικίνδυνο κομμάτι. Ε, θα πάρει όμως μια ένα μικρότερο κομμάτι του προπολογισμού, ανάλογα με το τι χρειάζεται, ενδεχομένως θα ε, προσθεθούν και κρατικά κονδύλια ε, και η ιδιωτική επένδυση θα γίνεται είτε παράλληλα είτε πάνω από αυτό. Ε, το στόχος του Ταμείου είναι να είναι καταλήτης για τις ιδιωτικές επενδύσεις και να αναλάβει κάποιο κίνδυνο, κίνδυνο που θα έχει σχέση με την ε, μακροπρόθεσμη κερδοφορία κάποιων σχεδίων τα οποία οι ιδιώτες επενδυτές ενδεχομένως διστάζουν να χρηματοδοτήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συνάδελφος Μούντι από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Thank you. Uh, yes, I just want... Σας ευχαριστώ σε σχέση με τις απαντήσεις όσον αφορά τον ορίζοντα 2020 και τις ε, επιπτώσεις που μπορούμε να έχουμε από το ότι ενδεχομένως να πάρουμε κάποια κονδύλια από τον τομέα της βασικής έρευνας. Κονδύλια τα οποία δεν πρόκειται όμως να αντικατασταθούν από τη νέα αυτή χρηματοδότηση η οποία προβλέπεται στα πλαίσια του EFSI. και φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή στερείται τη θεμελιώδη έρευνα από μια μελλοντική χρηματοδότηση. Αλλά ξέρετε ότι είναι έρευνα αυτή η οποία θα φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας, στην πρώτη γραμμή της καινοτομία. Νομίζω λοιπόν ότι μακροπρόθεσμα η δράση αυτή θα αποτελέσει τελικά αντικίνητρο όσον αφορά περαιτέρω επενδύσεις ή ακόμα μπορεί να οδηγήσει και σε αποβιομηχανοποίηση ορισμένων περιοχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ να πω τρία πράγματα όσον αφορά το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Πρώτον, από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφέ ότι θα έχουμε περισσότερα κονδύλια, περισσότερες πιστώσεις στους τομείς εκείνους που καλύπτει ορίζοντας 2020 μέσω του παράγοντα μόχλευσης που περιλαμβάνεται στο EFSI. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, επιδοτήσεις, μπορούν να χρηματοδοτήσουν κάποια έργα, αλλά υπάρχουν και έργα τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τον ιδιωτικό τομέα. Και ξέρω ότι υπάρχει μια σημαντική ανησυχία όσον αφορά αυτή τη μόχλευση επί 15, που ενδεχομένω να μην συνάδει με τα έργα τα οποία στο παρελθόν χρηματοδοτούνταν από επιδοτήσει. Ω προ αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είμαστε σαφείς. Αυτή η μόχλευση επί 15 έχει να κάνει με το σύνολο του χαρτοφυλακίου. Δεν αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή σε μία μόχλευση, σε ένα κριτήριο απέτηση μόχλευσης ανά project, ανά έργο. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων θα έχουμε γενικά μια μόχλευση της τάξης του 15, αλλά μπορούμε στη συνέχεια από το ένα project στο άλλο, από το ένα έργο στο άλλο, να έχουμε διαφορετικούς βαθμούς μόχλευσης. Αυτό το έχουμε δει και στο παρελθόν. Και θεωρούμε ότι θα καλυφθούν κατά αυτόν τον τρόπο πολλά προγράμματα τα οποία προβλέπονται αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα 2020. Προγράμματα τα οποία λάμβαναν επιδοτήσει στο παρελθόν. Κάτι ακόμα όσον αφορά το ζήτημα της προσθετικότητος. Είναι πολύ σημαντικό. Τα κονδύλια στα πλήσια του ΕΦΣΥ ουσιαστικά ανταποκρίνονται σε έργα τα οποία δεν θα βρίσκανε διαφορετική χρηματοδότηση. Αν το ΕΦΣΥ χρηματοδοτήσει έργα τα οποία θα χρηματοδοτήσει το ιδιωτικό τομέα, αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Δεν θέλουμε εμεί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε εμεί να προσελκύσουμε επιπλέον επενδύσει 315 δισεκατομμυρίων σε τριετή περίοδο και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις για τομείς οι οποίοι δεν θα χρηματοδοτούταν ούτως ή άλλως. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το επιπρόσθετο αυτό στοιχείο, ότι τα χρήματα δηλαδή θα καταλήξουν στα έργα εκείνα τα οποία έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Τζάνι που είναι μέλος και στις δύο επιτροπές και ΕΚΟΝ και ε, τώρα όμως σας αναλογεί ε, η Επιτροπή Οικονομικών. Σας ευχαριστώ. Τρία σημεία θέλω να θίξω. Πρώτον, μια διευκρίνηση όσον αφορά την απάντηση που δόθηκε στην ερώτηση παριθμών 4. Αν κατάλαβα κανά, το Ευρωπαϊκό αυτό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ουσιαστικά δεν θα χρησιμοποιεί μόνο τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά θα χρησιμοποιήσει επίσης και μέσω ομολόγων 60 δισεκατομμύρια σε περίοδο τριών ετών. Ποιο είναι το επιπλέον όμως χρέος το οποίο θα προκύψει για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεύτερον, όσον αφορά τις νέες επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι θέλει να προσελκύσει 315 ε, δισεκατομμύρια σε νέες επενδύσεις μέσω του ταμείου αυτού. Ελοχεύει όμως ο κίνδυνος αντί να έχουμε περισσότερες τελικά επενδύσεις, να βάλουμε κατά της δομής χρηματοδότησης των έργων που ήδη χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή με το παραδοσιακό σύστημα, όπως μπορεί να γίνει με τα project bonds. Ποιε είναι οι εγγυήσεις που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά μόνο για νέε επενδύσει. Και τρίτον, όσον αφορά του τρει πυλώνες στου οποίου αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε αντίθεση με τους δύο πρώτους ε, πυλώνες, ο τρίτος πυλώνας, ο οποίος προσελκύει ιδιωτικές επενδύσεις. Για τον τρίτο αυτό πυλώνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα του Ταμείου, διότι αυτή τη στιγμή δεν δίνεται κανένα μήνυμα προς τους ιδιώτες επενδυτές ότι πρόκειται να αλλάξει το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του νέου αυτού Ταμείου θα μπορούσε και για αυτό το σημείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι ακριβώς μπορεί να κάνει, προκειμένου να δώσει περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για τον τρίτο πυλώνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση παριθμών 4 και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη βαθμολογία της, είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει στα 3α διότι αυτό επιτρέπει τη φθηνή χρηματοδότηση των έργων. Υπό την έννοια αυτή, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων όντω θα αναλαμβάνει υψηλότερο κίνδυνο από ό,τι συνήθω η ΕΤΕ. Αλλά είναι προφανές ότι ο υψηλότερο κίνδυνο απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγύηση. Ε, Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί για να μην φυγεί ο βαθμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για μας είναι πολύ σημαντικό τα μεμονωμένα έργα τελικά ε, να ε, εποφεληθούν από την πολύ φτηνή χρηματοδότηση ε, της ΕΤΕ. Ε, σε σχέση με τον κίνδυνο αντικατάστασης φυσταμένων έργων, η προσθετικότητα είναι κάτι που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα βεβαιωθούμε ότι θα γίνει αυτό σε διάφορα επίπεδα. Πρώτον, η ανεξάρτητη επενδυτική κοινότητα παρακαλείται να μην ε, αναλαμβάνει έργα στα οποία δεν πιστεύει. Ε, θα υπάρξει μια επιτροπή που θα το ελέγχει διαχειριστική και θα υπάρχει και η λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στις ε, διάφορες εκθέσεις, στις οποίες θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να αναφερθούμε αργότερα. Για το τρίτο πυλώνα, όπως είπατε και εσείς, είναι ουσιαστικό το στοιχείο του πακέτου αυτού του επενδυτικού. Και για τους λόγους ακριβώς που αναφέρεται είναι τόσο κρίσιμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να κοιτάξει και να μελετήσει τι πρέπει να αλλάξει στο κανονιστικό πλαίσιο. Στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 αναφέραμε τέτοια στοιχεία για την ε, Ενεργειακή Ένωση, την Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών που προσπαθούμε να κάνουμε ε, προτάσεις για να μειωθούν τα ε, κανονιστικά εμπόδια έτσι ώστε να τονωθούν οι επενδύσεις στις ομίλους αυτούς. Ευχαριστώ. Ε, sorry, may I quickly come back on the first point? Μπορώ να επιστρέψω στο πρώτο σημείο ξανά λίγο. Δηλαδή, για να είμαστε σαφείς, όσον αφορά το επιπλέον αυτό χρέος που θα προκύψει για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είστε πεπισμένοι, είστε μια εγγύηση τελικά από, τις, από τους οίκους αξιολόγους ότι δεν πρόκειται να τροποποιήσουν το τριπλό α που έχει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι οίκοι αξιολόγησης εργάζονται μόνο και βαθμολογούν το τελικό προϊόν. Δεν επιτρέπεται καν ε, βάσει κοινοτικού δικαίου να κάνουν εκτιμήσεις πριν ολοκληρωθεί. Αλλά ε, έχουν πληροφόρηση, ε, δημοσιεύουν τα στοιχεία τους και λαμβάνεται υπόψη στην όλη χάραξη και σχεδιασμό του προγράμματος και του έργου να μην διακυβευτεί το τριπλό α. Ωραία, τηρήσατε τους χρόνους σας, γι' αυτό επιτρέπεται αυτή η ερωταπόκριση. Η κυρία Γκαρδία Σάβαλα από την Επιτροπή Προπολογισμών είναι επόμενη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτη μου ερώτηση έχει σχέση με το Ταμείο Εγγύσεων, το εγγυοδοτικό ταμείο το οποίο θα πρέπει να θεσπιστεί έτσι ώστε να λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Από πού βγήκε το νούμερο στόχος 50%. Γιατί αν το συγκρίνουμε με άλλα ταμεία παρόμοιων χαρακτηριστικών, όχι ίδια, σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε ε, μια τόσο σημαντική προστασία στο 50%. Από πού βγήκε ότι πρέπει η χρηματοδότηση να γίνει κατά 50% από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Εμεί όσοι. Ε, αυτό είναι μια ανησυχία, ε, διότι έτσι περικόπτονται πολύ και το ορίζοντα 2020 και το συνδέοντα στην Ευρώπη. δεύτερον, με αυτές τις περικοπές δεν καταλαβαίνω ακόμα πώς λειτουργεί το κριτήριο της προσθετικότητας. Δηλαδή, πώς είναι να κάποια σχέδια να είναι πρόσθετα όταν για να τα χρηματοδοτήσουμε περικόπτουμε από κονδύλια και γραμμές του προπολογισμού που είναι κανονικά αφιερωμένα και αφιερωμένες σε παρόμοια προγράμματα. Ασφαλώς ο στόχος είναι να έλξουμε ε, δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια αλλά ε, δεν πρόκειται για μια ε, δωρεάν ενίσχυση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Ε, υπάρχουν προγράμματα τα οποία ε, έχουν αμυγή κοινοτική χρηματοδότηση, υπάρχουν προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτεί ο ιδιωτικός και ο τομέα, αλλά το ταμείο αυτό αφορά αυτά που βρίσκονται ανάμεσα στα δύο. Ε, δεν είναι λογικό να κάνουμε μια απλή μεταφορά χρημάτων από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και μάλιστα σε τέτοιο ύψο προ την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να θέσει εφαρμογή αυτό το ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση, Πώ πώς υπολογίσαμε το στόχο 50%. Έχετε δίκιο. Είναι υψηλότερο αυτό το ποσοστό από ότι για άλλα ε, κατά μία παράδειγμα για την εξωτερική ε, εντολή. Για ποιο λόγο όμως. Ε, είναι η φύση του Ταμείου. Ε, το, το Ταμείο της Εξωτερικής Εντολής είναι, αφορά δάνεια σε χώρες. Εδώ μιλάμε για δάνειο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα δανείζει για συγκεκριμένα project. Επίσης, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναλάβει μεγαλύτερους κινδύνους Οπότε θα ήταν σόφρον να έχουμε ένα υψηλότερο ποσοστό. Ε, κάναμε ε, προσωμιώσεις ε, ενδεχόμενων ζημιών, ενδεχόμενων κερδών από τις δραστηριότητες του Ταμείου και το 50% ε, είναι στο, το κάτω όριο. Για την ακρίβεια, όχι το κάτω είναι ό,τι χρειάζεται. Ούτε υπερβολικά χαμηλό, ούτε υπερβολικά ψηλό. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε σίγουροι, επαρκώ σίγουροι ότι θα είναι ικανό και να προσθέσουμε και ένα μικρό ποσοστό έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον δεν θα χρειαστεί να αντλήσουμε περισσότερα κονδύλια από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Έτσι ώστε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να έχουμε ένα περιθώριο, ένα μαξιλαράκι. Τώρα, η προσθετικότητα. Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν κάποια project τα οποία μπορούν να χρηματοδοτούν μόνο με ε, δωρεάν ε, ενίσχυση, ε, επιδότηση δηλαδή, κάποια άλλα μόνο από τον ιδιωτικό το, τομέα από τα κράτη και το Ταμείο βρίσκεται, από, βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Ε, ο, γι' αυτό το, το λόγο προτεραιότητά μας εξακολουθούν να είναι επιδοτήσεις. Ε, αυτό που κάνουμε απλώς είναι ένα μικρό κομμάτι από αυτό το μετακινούμε στο, στο ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων και μάλιστα παίρνουμε λίγο από κάθε ε, δικαιούχο. Ε, εμείς εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι πρέπει να χρηματοδοθεί από την αγορά, να χρηματοδοτηθεί από την αγορά, ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, από αυτόν. Αλλά υπάρχει και ένα πεδίο ενδιάμεσο το οποίο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την αγορά, χρειάζεται να στήριχθει τουλάχιστον η πλευρά του κινδύνου του, έτσι ώστε να υλοποιηθούν αυτά τα project. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Βαμπρέμπτ από την Επιτροπή Βιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Αναφέρεται στην απάντησή σα στην ερώτηση του Ούντο Μπούλμαν, την πρώτη, ότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι πραγματικά κλειδί και στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Ταμείου στρατηγικών επενδύσεων. Αν δείτε την αιτιολογική σκέψη 14 στον κανονισμό του, στόχος είναι έργα που να έχουν υψηλή αξία για την κοινωνία και την ε, οικονομία, ιδιαίτερα έργα που προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, ανταγωνιστικότητα και μακροπρόθεσμη και μακροχρόνια μάλλον ανάπτυξη. Ωραία είναι όλα αυτά ως στόχοι, αλλά χτες ε, συζητήσαμε για τα ενεργειακά και πρέπει να ε, πετύχουμε τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μέλλον, ε, αβιώσιμες μεταφορές, ε, ενεργειακή απόδοση, αλλά εντάξει αυτό. Ποια είναι όμως η κοινωνική αξία και η βιωσιμότητα και πώς θα ληφθεί υπόψη. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να συμπεριφθούν και κριτήρια στον κανονισμό για να βεβαιωθούμε ότι τα έργα ανταποκρίνονται στους στόχους που ορίζει και σας ερωτώ, σε ποιο σημείο του κανονισμού θα συμπεριληφθούν αυτά τα κριτήρια για να μπορούν να κρίνονται ακριβώς και να εξετάζονται τα έργα ως προς την οικονομική τους ωφέλεια, την κοινωνική και τη βιωσιμότητα. Και ποια κριτήρια θα συμπεριλάβετε, αν συμπεριλάβετε. Για να συνδεθούν και να προσημειωθούν και σας παρακαλώ να μην δώσετε την ίδια απάντηση που δώσατε και στο έγγραφό σας, διότι δεν είναι αρκετή, δεν μας καλύπτει. Λέτε ότι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι να υπάρχει συμβατότητα με τις κοινοτικές πολιτικές. Εάν αυτό μόνο θέλετε, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Παρακαλώ, συμπληρώστε την απάντησή σας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Όντως, το εκτιμώντας 14 βρίσκουμε τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Καμία διαφωνία, όντως θα πρέπει το ΕΦΣΙ να στοχεύει στα έργα αυτά, όχι μόνο για έργα τα οποία βραχυπρόθεσμα μπορούν να ελοποιηθούν, αλλά για να πετύχουμε ακριβώς και αυτή την οικονομική, κοινωνική ωφέλεια και τη βιωσιμότητα στις οποίες αναφερθήκατε. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια δηλαδή της πρώτης κανονισμού έχουμε τη συμμετοχή και τη συμφωνία της EIB, ε της ΕΤΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έπειτα το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να θέσει κάποιες κατευθύνσεις. Εμείς θέλουμε προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαζόμαστε με τους συνομοθέτες για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ισορροπία ανάμεσα στους τρεις συμμετέχοντες αν οι συνομοθέτε θεωρούν ότι περισσότερα πράγματα θα πρέπει να ενταχθούν στον κανονισμό για να είναι πιο σαφή τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία αναφερθήκατε, τότε εμεί είμαστε διαλλακτικοί, μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σα για το πού μπορούν να περιληφθούν αυτά τα στοιχεία και πώς. Από τη δική μας πάντως την πλευρά θεωρούμε ότι ανταποκρινόμαστε μέσω της πρώτας αυτή τη στιγμή στους στόχους που μπορουν να περιληφθουν αυτα τα στοιχεια και πω απο τη δικη ενλοποιηθούν παντω την πλευρα θεωρουμε οτι ανταποκρινομαστε μεσω τη προταση αυτη τη στιγμη στου στοχου που αναφερθηκατε αρα εμεις δεν εντοπίζουμε κάπου κάποιο πρόβλημα. Τώρα πω θα αυτά στην πράξη. Πάλι έχουμε δύο επίπεδα εδώ πέρα. Το επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τα ζητήματα αυτά, αλλά παράλληλα θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που θα έχουν οι ίδιοι οι συνομοθέτε όσον αφορά τη λογοδοσία και όσον αφορά τη διαδικασία αναθεώρηση. Και το αναφέρω αυτό γιατί αν για οποιοδήποτε λόγο εσείς δεν είστε ικανοποιημένοι με την πορεία που ακολουθεί αυτό το ταμείο, υπάρχει ένας μηχανισμός υποβολής αναφορών και ένας μηχανισμός αναθεώρησης που θα μας επιτρέψει να λάβουμε υπόψη αυτές τις ανησυχίες. Μετά από 18 μήνες, μετά από 3 χρόνια γίνεται αναθεώρηση, Επίσης προβλέπεται στη συνέχεια ολοκληρωτική αναθεώρηση και ενδεχόμενη νέα υποβολή πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, Υπάρχουν τακτικοί μηχανισμοί για συστηματική αναθεώρηση και υποβολή αναφορών, έτσι ώστε όχι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και εσείς οι συνομοθέτες να μπορείτε να αποφαίνεστε για το αν κινείται σωστά ή όχι το Ταμείο αυτό. Ευχαριστώ από την Επιτροπή Μεταφορών, ο συνάδελφος Πίπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό τον καιρό ψάχνουμε εναλλακτική χρηματοδότηση και φαίνεται ότι το Συμβούλιο δεν διάκειται και τόσο αρνητικά απέναντι σε αυτό από ό,τι ακούω από τη χθεσινή συνεδρίαση. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη ε, για τη δεύτερη περίοδο, αν βγάλουμε τις χώρες συνοχής, ε, έχει μειωθεί σε 0,4 δις ε, από τα 2,7. Δηλαδή έχει πεθάνει το Connecting Europe Facility εκτός των χωρών συνοχής, επαναλαμβάνω. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα εξασφαλίσετε ότι τα κριτήρια που χρόνια ολόκληρα φτύσαμε αίμα για να διαπραγματευτούμε, η εθνική φάκελη, η διασυνοριακή ε, ε, μορφή μεταφορών, οι διάδρομοι, οι συνδυασμένες μεταφορές, όλα αυτά που πραγματικά τα έχουμε κατονομάσει συγκεκριμένα πώς θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων την επιβίωσή τους, γιατί τα νέα έργα έρχονται κατόπιν προτάσεων των κρατών μελών. Πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά και θα μεταφραστούν και θα ληφθούν υπόψη στο νέο επενδυτικό σχέδιο, που πραγματικά μας κόστησε πάρα πολύ για να το βάλουμε στο Connecting Euro. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να διευκρινίσω το εξή. Προτάσει για σχέδια μπορούν να προέρθουν από οποιονδήποτε. Οι ιδιώτε λοιπόν ενθαρρύνονται να υποβάλουν τέτοιου είδου προτάσεις. Δεν θα υπάρχει κάποιο φίλτρο έτσι ώστε να του απαγορευτεί. Δεν πιστεύω ότι το συνέοντα στην Ευρώπη ε, έχει καταργηθεί, που εξακολουθεί να είναι μία από τις προτεραιότητες ε, της Κομισιόν. Και το επιχείρημα είναι ίδιο με το αυτό του ορίζοντα 2020 ε, σε ό,τι φορά τα χρήματα που θα κατευθύνονται στα έργα. Εμείς προτείναμε να μην γίνουν μεταφορές μεταξύ τους. Όμως, ε, οι μεταφορές και οι, γενικότερα οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές ε, στο, στην ε, δραστηριότητα του Ταμείου. Οπότε εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι και για τον Ρίζοντα 2020 και για το Σύνοδο στην Ευρώπη τελικά περισσότερα χρήματα θα φτάσουν στους ενδεχόμενους δικαιούχους από ότι θα έφταναν χωρίς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Δεμάζη από την ε, Οικονομική Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε μια απάντηση δική μου ε, αναφέρεται ότι ε, θα υπάρξουν πολλαπλασιαστές ε, ε, από το κράτος ε, και το, το μεταφράζω αυτό ότι θα πρέπει να υπάρξουν μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις ιδιαίτερα στις χώρες της κρίσης και χρειάζεται μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση μεγαλύτερο ποσοστό ε, των κρατών μελών. Γιατί έχετε επιλέξει να ποντάρετε στη δημόσια προστασία ιδιωτών επενδυτών, ενώ υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και υπάρχουν και ομόλογα που μπορούν να αγοράσουμε εγγυημένα. Και επίσης, ποιος είναι ε, αυτός ο πολλαπλασιαστής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Υπάρχουν ιστορικά στοιχεία ε, που μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν χρησιμοποιείτε εσείς κανένα χρονολογικό. Και αυτοί οι πολλαπλασιαστές ε, εξαρτώνται πάρα πολύ και από το χρόνο και από την εκάστοτε συγκυρία. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα λοιπόν που έχετε χρησιμοποιήσει ε, και ε, θέλω να σας ρωτήσω και για τις ΔΙΤ, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού ε, τομέα. Λέει το Γερμανικό Ελεκτικό Συνέδριο ότι είναι πιο ακριβή αυτή η ιστορία γιατί θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι απαιτήσει των ιδιωτών για κέρδος. Γιατί επιλέγετε λοιπόν αυτό τη μορφή ΔΙΤ, γιατί είναι υπερχρεωμένα τα κράτη απαντάτε. Μα αυτό δεν είναι επιχείρημα ε, για να ακριβίνει περισσότερο το έργο, για να πληρώνουμε τον ιδιώτη και πώς ε, μπορείτε ε, να το δικαιολογήσετε αυτό με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που δεν εξαιρείται από εκεί κάποιες επενδύσεις των κρατών μελών αλλά όταν κερδίζουν οι ιδιώτες επενδυτές ξαφνικά αυτό γίνεται. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό μέσα στα πλαίσια που ισχύουν τα κανονιστικά. Ευχαριστώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα τρία αυτά σημεία. Στην πρότασή μας είμαστε σαφείς. Δεν έχουμε ως στόχο συγκεκριμένες χώρες, ε, δεν εστιάζουμε σε συγκεκριμένες χώρες. Ασφαλώς και ο πολλαπλασιαστής θα είναι διαφορετικός για κάθε χώρα. Αλλά επιθυμία μας ήταν να αποφύγουμε να εστιάσουμε γεωγραφικά ή θεματικά. Για ένα λόγο. Όπως λέτε και εσείς, η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο τη συμμετοχή των ιδιωτών μέσω παραγωγικών επενδύσεων. Αν εντοπίζαμε τη δράση μας θεματικά ή γεωγραφικά, πάντοτε θα ανησυχούσαμε για το ότι ενδεχομένως θα επιλέγαμε έργα τα οποία δεν είναι βιώσιμα, ε, θα ότι δηλαδή θα τα επιλέγαμε επειδή χρειάζεται οπωσδήποτε να δοθεί ένα συγκεκριμένο ποσό σε μια χώρα, σε ένα τομέα. Τώρα, ομόλογα που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συγγνώμη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα εκδώσει ομόλογα ασφαλώ, αλλά δεν ξέρω αν θα ήταν νόμιμο να τα εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχω την εντύπωση πω όχι. Σε ό,τι αφορά τη μόχλευση και το χρονικό διάστημα, ε, το αν θα είναι έξι, ε, αν, αν, βάλουμε 6 μήνες, 3 χρόνια, 5 χρόνια, ε, ως διάρκεια, τότε η, το ποσό της μόχλευσης ε, ε, διαφέρει. Τώρα, αυτό το 15, αποκαλυψιαστής 15, έχει σχέση όχι τόσο με μια συγκεκριμένη περίοδο για ένα συγκεκριμένο μέσο, χρηματοδοτικό μέσο. Ξετάσαμε το παρελθόν της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και την εμπειρία της με χρηματοδοτικά όργανα, αλλά χρησιμο, ε, λάβαμε υπόψη και γενικότερα την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο στοιχείο που μπήκε εκεί, στον πολλαπλασιαστή, είναι το, η δουλειά που έχουμε κάνει εμείς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, για το τι θα κάνει, ποιες θα είναι οι δραστηριότητε του Ταμείου. Μπορείτε να μου πείτε πιο συγκεκριμένα. Ε, ε εμείς είδαμε, ε, λάβουμε υπόψη μας περίπου τρία χρόνια για το Ταμείο. Ζητήσαμε 350 δισεκατομμύρια προς τον επενδύσεων για τρία χρόνια. 315 δισεκατομμύρια προς τον επενδύσεων για τρία χρόνια. Οπότε για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τα έχουμε υπολογίσαμε τον ε, πολλαπλασιαστή. Τώρα, για το τρίτο ερώτημα σας δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα διορθώστε με αν κάνω λάθος, τα κράτη-μέλη θα συνεισφέρουν ε, και η συνεισφορά τους θα αξιολογηθεί με διάφορους τρόπους, ανάλογα το πού θα συνεισφέρουν. Εμείς ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ε, συνεισφέρουν σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στατικών Επενδύσεων. Αυτό είναι προς συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οπότε ε, με αυτόν τον τρόπο ε, θα διασφαλίζεται η ε, μεταχείριση, ιδιαίτερη μεταχείριση, προνομιακή μεταχείριση. Τώρα, οι επένδυσεις, οι συνεισφορές σε επίπεδο έργου δεν έχουν τέτοιου είδους μεταχείριση. Πάντοτε υποστηρίζαμε ότι θα πρέπει ε, να υπάρχει μια, να μην οδηγηθούμε σε, υπερβολικά, σε υπερβολικό δανεισμό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνονται παραγωγικές επενδύσεις αλλά χωρίς υπερβολικό δανεισμό. Μάλιστα. Σας είπα ότι είναι πάρα πολύ λεπτή η κατανομή ε, ανάμεσα στις διάφορες επιτροπές ο κατάλογος αγορητών. Ο κύριος Έλερ έχει το λόγο, γιατί έχουμε και ε, εισηγητές και σκιώδες. Τις ερωτήσεις έχω. Ερώτηση πρώτη. Ο Επίτροπος Κατάινεν επανειλημμένα έχει τονίσει ότι η ε, ε, τα δάνεια ε, έχουν ένα πολλαπλασιαστή 15 και στον ορίζοντα 2020 για κάθε δισεκατομμύριο που βάζετε παίρνετε 13. τι ισχύει, ισχύει ο υπολογισμός στο ορίζοντα ε, το ταμείο έχει πολλαπλασιαστεί αλλά οι επιδοτήσει όχι, ε, όπως λέει ο κύριος Κατάινεν, ποιος έχει δίκιο. Και επίσης λέτε δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιφερειακές πλατφόρμες. Ε, με το σχέδιο για το Ταμείο Επενδύσεων που δημοσιεύτηκε, όχι δεν δημοσιεύτηκε, απλώ διέρευσε. Contributions from third parties από τρίτη τους λοιπόν οι συνεισφορές θα μπορούν να καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές για ε, διάφορες συμφωνίες ε, ε, πολλαπλών προγραμμάτων. Αυτό είναι αντίφαση. Εγώ δεν θέλω να το αξιολογήσω, ούτε λέω ότι είναι αυτή μια εισαγωγή στα ευρωομόλογα, απλώς να μου πείτε τι εννοείται και τι λέει το νομοθετικό κείμενο και τι είναι τελικά οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είχε νόημα, πώς το βλέπετε τώρα, για λόγους πρακτικούς και ε, εφαρμοστικούς ε, δεν μπορούμε ε, να αλλάξουμε τώρα τα ισχύοντα για τον προπολογισμό και θέλετε να πάρετε χρήματα από το ΣΕΦ και από το ορίζοντα για να τα δώσετε σε αυτό το ταμείο. Ε, μπορεί να γίνει αυτό έμπροστο βαρέ, μετά να γίνει μια ενδιάμεση ε, αξιολόγηση του πολιετέ δημοσιονομικού πλαισίου και να ξέρουμε πόσα λεφτά έχουμε. Γιατί ο ορίζον αυτή τη στιγμή δεν χρηματοδοτείται από τον ορίζοντα, διότι ε, δεν έχει χρήματα καθόλου, τα παίρνετε απαλού. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα εμπροστοβαρό κάποια χρήματα και στην ενδιάμεση αναθεώρηση να φροντίσουμε να υπάρχει μια γερή χρηματοδότηση για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Τρίτη ερώτηση. Γιατί μιλάτε για ε, στη 15 όταν όλες οι ε, κρατικές ε, τράπεζες ε, επενδύσεων και αναπτυξιακές δήλωσαν και ο ίδιος ο Κατάινεν ότι δεν θέλει να έχει private equity funds μία, αλλά μόνο από τα 8 δισεκατομμύρια ε, που υπάρχουν ως εγγύηση και οι υπόλοιπε εγγύησει θα έρθουν μόνο από τα 18 δισεκατομμύρια των εγγύησεων του προπολογισμού. Δεν ξέρω πώς τα υπολογίζετε αυτά, όλο αντιφάσει είναι. Θα δημιουργήσετε ένα νέο ε, εργαλείο εγγύησεων, δεν λέω ότι είναι λάθος, αλλά πού τα βρήκαμε τα 315 για private equities. Thank you. There were four questions, which I will take three and then pass to one ερωτήσεις σας ετέθησαν. Κοιτάξτε, οι προβλέψεις αυτές ε, δεν είναι σωστές. Σε ένα από το ερώτημα που μας ετέθηκε, απαντήσαμε χθε, ε, είπαμε ότι αυτή είναι ακριβώς η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι ότι οι επιδοτήσεις έχουν μηδενική μόχλευση, έχουν πολύ χαμηλή μόχλευση, αυτό είπαμε. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι επιδόματα δεν έχουν μόχλευση. Απλώς η μόχλευση αυτή είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή που προβλέπεται για άλλα χρηματοδοτικά μέσα, όσον αφορά τις περιφερειακές πλατφόρμες. Θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γραπτός λέει στο σχέδιο προϋπολογισμού για τον ορίζον 2020 ε, ότι ένα δισεκατομμύριο θα αποφέρει 13. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει για τον ορίζοντα ότι η μόχλευση είναι 13. Ισχύει ή δεν ισχύει. Αληθεύει ή όχι. Εγώ αυτό ρώτησα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη αν προκάλεσα σύγχυση. Αυτή η μόχλευση ευχαριστω και ζητω συγγνωμη προκαλεσα συγχυση αυτη η μοχλευση επι 13 έχει να κάνει με τα χρηματοδοτικά μέσα συν τις επιδοτήσεις για τον ορίζοντα 2020. Αν τα συνδυάσετε και τα δύο, τότε καταλήγετε σε αυτό το ποσό το οποίο αναφέρατε. Συγγνώμη αν προκαλέσαμε κάποια σύγχυση με την πρότασή μας. Όσον αφορά τώρα τις περιφερειακές πλατφόρμες και την περιφερειακή κατανομή πιστώσεων, πάλι μπορεί να μην είναι Αυτό το οποίο λέμε στην πρότασή μας είναι ότι δεν προβλέπεται περιφερειακή κατανομή από τον ΕΦΣΙ. Δεν λέμε ότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν περιφερειακές πλατφόρμες, απλώς δεν πρόκειται να έχουμε συγκεκριμένες πιστώσεις για συγκεκριμένους τομείς και συγκεκριμένες περιφέρειες στα πλαίσια του ΕΦΣΙ. Τα κράτη-μέλη, οι ιδιωτικές εταιρείες, όποιος το επιθυμεί, μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες πλατφόρμες και να χρησιμοποιήσουν κονδύλια από το ΕΦΣΙ και αν η Επιτροπή Επενδύσεων αποφασίσει στη συνέχεια ότι αξίζει να υποστηρίξει ο ΕΦΣΙ μια τέτοια επένδυση, τότε μπορεί να γίνει. Μπορεί να ληφθεί υπόψη δηλαδή η περιφερειακή αυτή συνιστόσα. Πάντω δεν πρόκειται εξ αρχή να έχουμε ω γνώμονα αυτή την περιφερειακή κατανομή των πιστώσεων. Δεν απαντάω αυτή τη στιγμή στην τρίτη ερώτηση να πω για την εγγύηση των 16 δισεκατομμυρίων. Πολύ φοβάμαι ότι προκαλέσαμε μία σύγχυση ουσιαστικά είναι το 100% των 16 δισεκατομμυρίων, ενώ τα 8 δισεκατομμύρια χρησιμοποιούνται για την ε, προστασία των προπολογισμών από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει αυτών των 16 δισεκατομμυρίων. Αναφερόμαστε λοιπόν στην εγγύηση των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εγγύηση για τις επενδύσεις αυτές. Τώρα, αν μπορεί να γίνει προς το βαρύς χρηματοδότηση στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, να δώσω το λόγο στον Αντουάν. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το είπαμε ήδη. Υπάρχει και το ζήτημα της πολιτικής σκοπιμότητας και δυνατότητας υλοποίησης του σχεδίου αυτού. Προφανώς πρέπει να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη καθώς επίσης και την τόνωση των θέσεων απασχόλησης. Πρέπει λοιπόν εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσουμε τις προτεραιότητες αυτές και γι' αυτό τον λόγο τα τρία θεσμικά όργανα είπαν ότι μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, να έχει εγκριθεί αυτή η πρόταση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει μέχρι τα μέσα του 2015 να έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά και για όλα τα προγράμματα τα οποία εντάσσονται αυτή τη στιγμή στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν εμείς τώρα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μέσω του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, τότε ελοχεύει ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα τα οποία δεν θα καταφέρουμε να διευθετήσουμε στο χρονοδιάγραμμα αυτό το οποίο έχουμε θέσει για τον ΕΦΣΥ, αλλά και στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του δημοσιονομικού πλαισίου. Μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτησή μου. Κοιτάξτε κύριε Έλερ, ε, ε, εντάξει, ήμουν αρκετά γενναιόδωρος με το χρόνο γόρευσης και έχω ακόμα 8 συναδέλφους, ζητώ συγγνώμη. Επόμενος συνάδελφος, ο κύριος Τσεχόφσκι από την Επιτροπή Προπολογισμών και παραδίδω και την Προεδρία στον συνάδελφο Γκολτιέρη. Ευχαριστώ. Έχω ε, εργαστή στην έρευνα και την κοινοτομία για αρκετό καιρό και έχω, μια, ε, έχω την εξή ερώτηση. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει μια εγγύηση του 10% του προϋπολογισμού, γιατί πιστεύετε ότι αυτό θα δώσει κίνητρο στους ιδιώτες επενδυτές να προσθέσουν τη δική τους συνεισφορά. Διάβασα την πρότασή σας και λέτε ότι θα χρηματοδοτείτε έργα τον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Εγώ προέρχομαι από την Κεντρική Ευρώπη και δυσκολευόμαστε να απορροφήσουμε τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Γιατί πιστεύετε ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν επιπλέον σχέδια. Εσείς λέτε τώρα βέβαια ότι θα πρόκειται για σχέδια, τεχνολογία, λέιζερ, τις μεταφορές, τις υποδομές κλπ. Πιστεύετε ότι ε, θα επιτευχθούν οι πρόσθετες επενδύσεις ε, ε, στις οποίες αναφέρεστε και θα, προσκληθεί θα το ιδιωτικό κεφάλαιο που είναι απαραίτητο. Επιτροπή. Ε, δύο ερωτήσεις. Γιατί πιστεύουμε ότι η εγγύηση του 10% θα αποτελέσει κίνητρο για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Η εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν θα εγγυηθούμε τίποτα για τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς θα εγγυηθούμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συλλέξει πρόσθετα κονδύλια για να υποστηρίξει τα σχέδια, τα έργα. Το ποσοστό είναι πάνω από 10%. Εξαρτάται από το έργο, αλλά από ό,τι είδα σε μια αιτιολογική σκέψη, θα φτάσει περίπου στα 60 δισεκατομμύρια. Τα 60 δισεκατομμύρια θα επενδυθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να αποτελέσουν μαγιά, καταλήτη, έτσι ώστε να προσελκυστούν ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο τώρα. Το βασικό στοιχείο εδώ είναι η προσθετικότητα. Ε, εστιάζουμε σε έργα που δεν μπορεί να τα υλοποιήσει από μόνο του ιδιωτικό τομέα εξαιτία του γεγονότο ότι υπάρχουν εγγενεί κίνδυνοι. Ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος είναι αυτός ο οποίος πολλές φορές ε, ε, αποτελεί αντικίνητρο για του ιδιώτε επενδυτέ. Για παράδειγμα, πολλοί από αυτού μπορούν να δουν ένα πολύ καλό έργο, αλλά δεν θέλουν να αναλάβουν κίνδυνο για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Και μιλούμε ακριβώ για τέτοιου είδου σχέδια, τα οποία αργότερα οι επενδυτέ δεν μπορούν να τα πουλήσουν εύκολα, να τα εμπορευτούν. Οπότε αυτή η εγγύηση θα αποτελέσει καταλήτη για τον ιδιωτικό τομέα. Για το δεύτερο σας ερώτημα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στον τομέα της έρευνας είναι και πάλι να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια. Ορισμένους από τους τομείς, ε, για παράδειγμα, που παλιότερα ε, το μέσω επιδοτήσεων, αλλά και άλλους που χρειάζονται ιδιωτικά κεφάλαια. Ορισμένοι τομείς έχουν ε, δυσκολευτεί να απορροφήσουν τα περιφερειακά κονδύλια που βρίσκονται στη διάθεσή τους. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι η ιδιωτική έρευνα και ανάπτυξη. Το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων θα επιτρέψει ε, να ε, διευκολυνθεί η ιδιωτική επένδυση σε αυτούς τους τομείς με τρόπους που δεν γινόταν παλιά. Εμείς το βλέπουμε ως πρόσθετο, όχι ως ανταγωνιστικό των περιφερειακών ταμείων, των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης. Θέλουμε το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να συμπληρώσει τα περιφερειακά ταμεία σε κάτι λίγο διαφορετικό. Thank you. Now Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέρμερ από την Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χωρίς μεγάλη εισαγωγή θέλω να κάνω κι εγώ σημαντικές για μένα ερωτήσεις γίνεται λόγος για αυτή τη χρηματοδότηση που θα έχει λέει τόσο καταπληκτικά αποτελέσματα. Τότε θα σας παρακαλούσα να μου πείτε ε, ποια είναι η διάρκεια αυτών των χρηματοδοτήσεων, για ποιο χρονικό διάστημα μιλούμε. Γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και κάποιες απώλειες. Αυτές οι απώλειες πότε αναμένονται. Ποιος το καθορίζει, ποιος το διαπιστώνει και μήπως υπάρχουν φόβοι και ανησυχίες ε, όταν είναι περιορισμένα τα κρατικά χρήματα και οι κρατικές εγγύησεις, μετά μήπως κινδυνεύουμε να χρηματοδοτούμε μέσα που δεν είναι εγγυημένα και τελικά να πει ε, ο ένας ή ο άλλος ότι τώρα θα πρέπει να κάνουμε τις απώλειές μας γιατί δεν θα μας δώσουν κρατικές εγγύησεις. Και οι τράπεζες πώς θα υπολογίζουν τα κέρδη και τις ζημίες τους. Υπάρχει διακίνδυνο να παραμείνουν ε, τα κέρδη ε, στους επενδυτές και ε, οι ζημίες στους φορολογουμένους. Γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό όταν σώσαμε τράπεζες και όταν σώσαμε χώρες. Παράδειγμα την Ελλάδα. Και ε, αν είναι μόνο 16 δισεκατομμύρια ε, από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, μήπως θα πρέπει να φροντίσουμε το σύνολο του ποσού αυτό να προστατεύεται κάπως γιατί μπορεί να, ε, να χαθεί τον προϋπολογισμό. Παρακαλώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. the two... Σας ευχαριστώ για τις δυο σας ερωτήσεις. Η διάρκεια της χρηματοδότησης πρώτον. Πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό το οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 315 δισεκατομμύρια με τη μορφή επενδύσεων μέσα σε τρία χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της τριετούς περίοδου εξαφανίζεται η εγγύηση. Η εγγύηση θα υφίσταται για όλη τη διάρκεια του έργου αν είναι ένα έργο 5-6 ετών, τότε η εγγύηση θα το συνοδεύει για 5-6 χρόνια. Αν διαρκέσει το σχέδιο, το έργο αυτό 30 χρόνια, ανάλογη θα είναι και η διάρκεια της εγγύησης. Αλλά δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μπροστοβαρή χρηματοδότηση των απολειών. Ακριβώς επειδή η εγγύηση θα υπάρχει καθ' τη διάρκεια του έργου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να προσελκύσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Και είναι ακριβώς αυτός ο, το μακροπρόθεσμο αυτό κίνδυνο που θέλει να αποφύγει ο ιδιωτικό τομέας, που δεν θα μπορούσαμε εμείς να καταργήσουμε την εγγύηση. Τώρα, τι γίνεται με, τις, με τα κέρδη και τις ζημίες και ποια είναι η σχέση με τι τράπεζε. Για εμά το ερώτημα δεν τόσο πολύ ποια είναι τα κέρδη και ζημίες των τραπεζών, αλλά των έργων αυτών καθ' αυτών. Οι τράπεζε θα κερδοφορήσουν αν κερδοφορήσουν και τα ίδια τα έργα. Το αντίστροφο επίση θα συμβεί αν έχουμε ζημία σε ένα έργο, θα ζημιωθεί και η τράπεζα. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές και απόκληση κινδύνου, ιδίως με το σύστημα παρακολούθησης το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργείται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπου έχουμε καλύτερο έλεγχο κερδών και ζημιών. Όσον αφορά τώρα τις τράπεζες, οι τράπεζες μπορούν καταρχάς να επενδύσουν σε ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα οποία για να τα χρηματοδοτήσει θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εκδώσει περίπου 60 δισεκατομμύρια σε ομόλογα. Αυτό για το σύνολο του ισολογισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οπότε ακόμα και αν υπάρχει ζημία ή απώλεια σε ένα έργο δεν πρόκειται να επηρεαστεί κάποια τράπεζα, ακριβώς επειδή θα προστατεύονται και οι τράπεζε ή οποιοδήποτε άλλο ιδιώτη μπορούν να συμμετέχουν και κατά έργο, αναπερίπτωση δηλαδή. Φαντάζομαι ότι στα πλαίσια του CRD, την οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει γνωρίζετε ότι ακριβώς προβλέπουμε ότι οι τράπεζες δεν θα εκτίθενται σε πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ακριβώ για να καταφέρουμε να προστατεύσουμε αυτά τα δημόσια κονδύλια στα οποία αναφερθήκατε. Κύριε από την Επιτροπή ε, Υπολογισμού, όχι, κυρία Αγιάλα Σέντερ από τις μεταφορές προηγουμένω. Πρώτον, προ την Κομισιόν η εξή ερώτηση. Πριν φτάσουμε στην απόφαση περικοπής προγραμμάτων που τα είχαμε σχεδιάσει, υιοθετήσει κλπ. Σκεφτήκατε και το που θα μπορούσατε ενδεχομένω να βρείτε τα ίδια χρήματα, 8 δις, δεν ξέρω, 16, από άλλες πηγές του προϋπολογισμού. Που, χρήματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ταμείο για την ευελιξία, αποθεματικό κλπ. κλπ. Μπορείτε να μου πείτε τι, τι νούμερα είχε βγάλει αυτή η μελέτη. Δεύτερον, εγώ είμαι από τις μεταφορές. Τι σας κάνει να πιστεύετε, όπως είπατε πριν από λίγο, ότι θα έχουμε καλύτερα, πιο κερδοφόρα ε, προγράμματα, σχέδια, έργα από ό,τι τις ε, ε, στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό που βλέπω εγώ είναι ομόλογα για την για τη χρηματοδότηση αυτοκινητοδρόμων. Ε, αντίθετα όμως, στο συνδέοντας την Ευρώπη είχαμε και τους ιδιοδρόμους και τις πλωτές οδούς. Τώρα, ε, χώρες με πλεόνασμα και με έλλειμμα. Εσείς λέτε ότι θα συμμετάσχουν όλα τα κράτη-μέλη. Τι κίνητρο θα τους δώσετε. Τι κίνητρο θα δώσετε στις χώρες που έχουν ελλείμματα. Γιατί αυτοί θα το βλέπουν ως ε, δώρο μόνο για τους ε, πλεονασματικούς. Ε, μετά, στην ε, Επιτροπή των ε, Επενδυτών δεν ε, έχουν λόγο ιδιώτες. Τε, τέλος, γιατί εμείς θα χρηματοδοτούμε το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που θα ασχολείται με αυτό το ταμείο. Δεν έχουν χρήματα ούτε καν να πληρώνουν τους εμπειρογνώμονές τους. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλές ερωτήσεις κάνατε. Θα απαντήσω σε μερικές εγώ και σε άλλες, ε, άλλοι συνάδελφοι ε, που μπορούν να σας δουν πιο λεπτομερείς απαντήσεις από εμένα. Γιατί μας κάνει να πιστεύουμε ότι τα έργα ε, αυτά είναι πιο κερδοφόρα στο ΕΦΣΙ από ότι στο Συνδέοντας Ευρώπη. Δεν είναι εκεί το θέμα. Μπορεί και στην διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη να υπάρχουν πολύ κερδοφόρα έργα. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αντιφατικό ή ανταγωνιστικό. Ο ιδιωτικό τομέα αναγνωρίζει ένα έργο ότι συμφέρει, αλλά δεν είναι πρόθυμος να αναλάβει το ρίσκο. Και για να ξεκινήσει ένα έργο χρειάζεται μια μαγιά, μια επιδότηση και μετά για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί πλήρως πρέπει να βρεθούν τα χρήματα παλού. Αυτό προσπαθούμε να βρούμε εμείς στη χρυσή τομή, ε, ε, να δοθεί ένα κίνητρο στον ιδιωτικό τομέα να μπει και να τον βοηθήσουμε εμείς να δρομολογηθεί το έργο με την υποστήριξη του Ταμείου Στατηγικών Επενδύσεων. Ε, τώρα για τις χώρες ε, τις λιματικές και τις πλεονασματικές και τι κίνητρα μπορούν να τους δοθούν στις πρώτες. Από πλευράς μας είναι πολλά τα κίνητρα ανεξαρτήτως ε, του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για δημόσιες επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις δεν θα πρέπει να γίνονται μόνο μέσω του Ταμείου αυτού, ούτε θα πρέπει εμείς να το ενθαρρύνουμε κάτι τέτοιο. Πολλές χώρες εξέφρασαν, δήλωσαν προθυμία μάλλον στον τύπο, σε επίπεδο κράτους μέλους και σε επίπεδο περιφερειακό. Αυτό δεν εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα τους μεταχειριστούν, αλλά θέλουν να προσελκύσουν τα χρήματα στη χώρα τους. Τουλάχιστον αυτά διαβάζουμε από τον τύπο ότι έτσι θέλουν να μπουν τα κράτη-μέλη στο ΕΦΣΥ. Βεβαίω υπάρχουν πολλά κίνητρα για να επενδύσει κανείς ε, στη χώρα του για την οικονομία. Τώρα, το κόστος του προσωπικού, πριν δώσω το λόγο σε άλλους συναδέλφους. Το καταστατικό ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, προβλέπει και σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρωτόκολλο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επιδήσεων χρεώνει τις παροχές ε, και αυτό χρηματοδοτείται ε, κάθε έργο. Γι' αυτό είναι πολλά τα έργα για να επιμεριστεί το κόστος. Δεν είναι κόστος του προσωπικού. Δεν πληρώνει ο κοινοτικό προπολογισμό, δηλαδή του υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μια ακόμα ερώτηση νομίζω για ένα σενάριο χρηματοδότησης. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, το σενάριο χρηματοδότηση το οποίο έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν εξετάσαμε και εναλλακτικέ. Προφανώ το εξετάσαμε πολύ προσεκτικά η βασική υπόθεση, το βασικό σενάριο ήταν ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνει χωρίς να ανοίξει το δημοσιονομικό πλαίσιο εκ νέου, χωρίς δηλαδή να αναθεωρηθεί το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Διαφορετικά δεν θα ήταν το σχέδιο αυτό συμβατό με τον γενικότερο στόχο να προχωρήσουμε γρήγορα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν έχουμε αυτή την αλλακτική αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου λιγοστεύουν οι εναλλακτικέ. Βασικά, για να εγγυηθεί κανεί τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, πρέπει να κάνει ανακατομή, ανακατονομή των προγραμμάτων στο κεφάλαιο 1α, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το περιθώριο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του 1α και η μερική χρήση του γενικού περιθωρίου για τις πληρωμές αλλά και την άλυψη υποχρεώσεων. Αυτές είναι οι εναλλακτικέ. Βάσει λοιπόν αφού του πλαισίου έπρεπε να εργαστούμε, και στα πλαίσια του κεφαλαίου Α προσπαθήσαμε να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες ανακατανομής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να δούμε αν υπήρχαν κάποια προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν κατά πολύ, για παράδειγμα, αν μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια, δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να καταστρέψουμε προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν μόνο κάποιες χιλιάδες ευρώ. Προφανώς Εξετάσαμε βέβαια και την περίπτωση προγραμμάτων που θα μπορούσαν να μεταφέρουν επιστώσεις από κάποιους τομείς πολιτικής που έχουν πάνω κάτω τους ίδιους στόχους με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Έτσι καταλήξαμε λοιπόν στο σενάριο το οποίο περιλαμβάνει το ΣΕΦ και τον ορίζοντα 2020 και το κόσμο επίσης το εξετάσαμε, αλλά στα πλαίσια του κόσμου έχουμε άνω του 60% των πιστώσεων του ήδη δεσμευμένα μέσω άλλων χρηματοδοτικών μέσων. Το να πάρουμε περισσότερα λοιπόν, περισσότερε πιστώσει από το κόσμο δεν θα ήταν ρεαλιστικό και λάβαμε γι' αυτό υπόψη επίση και το κριτήριο τη προσθετικότητα. Sí, eh, solamente Δεν μου απαντήσατε ε, στο ερώτημα που σας έθεσα. Μιλούσα για τα χρήματα του προβλησμού που δεν χρησιμοποιούνται, για το αποθεματικό της ευελιξίας, δηλαδή το μαξιλάρι που υπάρχει και δεν έχει καμία σχέση με το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό το οποίο ετησίως ε, ε απομένει στον προπολογισμό και δεν το χρησιμοποιούμε ή δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Ε, για παράδειγμα, τους πόρους ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. υπάρχουν χρήματα τα οποία παραμένουν αχρησιμοποιητά στο τέλος κάθε ε, οικονομικού έτου, και επιστρέφονται δεν ξέρω πού ακριβώς, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όμως. Δεύτερον, σε, σε ό,τι αφορά τα, αυτά τα έργα τα οποία περιμένουν να χρηματοδοτηθούν, θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα-δυο παραδείγματα τέτοιου είδους έργα που δεν είναι αυτοκινητόδρομοι με διόδια, αλλά είναι τέτοιου είδους έργα τα οποία περιγράφεται. Great. Commission, yes. Να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, για τις μη χρησιμοποιούμενες πιστώσεις, ναι και όχι. Δεν μπορούμε εξ αρχής να δημιουργήσουμε μια τόσο μεγαλεπίβολη πρωτοβουλία με τόσα πολλά εμπλεκόμενα έργα χωρίς να γνωρίζουμε ότι θα έχουμε μόνιμη χρηματοδότηση για μεγάλο χρονικό διάστημα με συγκεκριμένη απόδοση επενδύσεων. Εξ αρχής έπρεπε να είμαστε σίγουροι να έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των έργων. Τώρα, το περιθώριο για τις υποχρεώσεις και το περιθώριο για τις πληρωμές είναι κάτι το οποίο είπαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να μετακινήσουμε, να μεταφέρουμε επιστώσεις από προηγούμενα έτη σε επόμενα έτη στα πλαίσια πάντα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δηλαδή, προφανώ το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο είχε ήδη αυτή την ευελιξία προτού εγκριθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και συνεχίζουμε να εκμεταλλευόμαστε τη δυνατότητα αυτή και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ευχαριστώ, ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ρωτήσεις θέλω να κάνω, πολύ απλές και άμεσες, αλλά ουσιαστικές για μένα. Πρώτον, ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι η επιλογή αυτών που θα στελεχώσουν την επιτροπή αυτή. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη καθώς επίσης και ανεξαρτησία της Επιτροπής αυτής των επενδύσεων, ότι οι άνθρωποι αυτοί όντως γνωρίζουν τον τομέα αυτό, ότι μπορούν όντως να συμβάλλουν με έργα τα οποία δεν θα έχουν μόνο πολιτικό χρώμα, δεν θα απαγορεύονται από τα λόπια, αλλά θα έχουν και κάποιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, τα 57 δισεκατομμύρια που θα δώσετε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πώς ακριβώς θα τα δώσετε, κυρίως σε νέες επιχειρήσεις startup, για παράδειγμα, που προωθούν καινοτόμα έργα. Ξέρετε ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν καταφέρουν να βρουν χρηματοδότηση για τα έργα τους, ακριβώς επειδή υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο κινδύνου πολλές φορές. Αλλά είναι αυτές οι επιχειρήσεις οι μικρές οι οποίες προωθούν περισσότερο την καινοτομία. Πώς θα βοηθήσετε τις καινοτόμες νέες επιχειρήσεις. Thank you. Two Ευχαριστώ. Δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Η επιλογή των μελών της επενδυτικής κοινότητας είναι, όπως είπατε, πάρα πολύ σημαντική. Είναι κρίσιμη, ακριβώς για να αποφευθεί η κατάσταση στην οποία αναφέρατε. Σε σχέση με αυτό, η πρόταση ε, θα διαμορφωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά ε, μετά την έκδοση της απόφασης είδαμε ε, ότι ε, υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την Επιτροπή Επενδύσεων. Εμείς θέλουμε να παραμένει απολύτως ανεξάρτητη η επενδυτική κοινότητα, γιατί σε αυτό βασίζεται. Συγγνώμη, Επιτροπή Επενδύσεων. Set 75 εκατομμύρια έχουν αφαιθεί στην άκρη 75 δις, συγγνώμη, ε, για τις εταιρείε αυτές και είναι πάρα πολύ σαφής η προσέγγιση μας ε, ως προς την προσθετικότητα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν πολλά έργα, ε, άλλα έχουν να κάνουν με το χρέος και άλλα με την ιδιωτική χρηματοδότηση. Ε, ξέρουμε ότι κάθε προσπάθεια χρειάζεται ξεχωριστή χρηματοδότηση, στοχευμένη, ανάλογα με την μικρομεσαία επιχείρηση. Ε, οι νεοφυείς, οι πάρα πολλοί καινοτόμες νέες επιχειρήσεις, ακριβώς αυτό χρειάζονται. Και αυτό που θέλουμε να βεβαιωθούμε είναι ότι υπάρχει επιπλέον προσθετικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now, next speaker is Maragall from the Budget Committee. Maragall από την Επιτροπή Προπολογισμών. Ένα μόνο σχόλιο σε ό,τι αφορά τους ε, όρους και τις προϋποθέσεις ε, για κάθε ένα από τα παιδιά του ΕΦΣΥ. Ε, είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι θα πρέπει να οριστούν με απόλυτη ακρίβεια και με το ελάχιστο, την ελάχιστη δυνατή δυνατότητα ερμηνείας τους. Οπότε έχω τρεις ερωτήσεις, πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, σύμφωνη η Κομισιόν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δίδεται ενίσχυση ή ως ενίσχυση ή ως εγγύηση ε, ακίνητο του κράτους. Επίσης δεν θα πρέπει να ζητείτε, να απαιτείτε παροχή υπηρεσιών, κρατικών υπηρεσιών. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να δίδονται εκ των προτέρων ποσοστώσεις, εδαφικές ποσοστώσεις. Συμφωνείτε ότι το Ταμείο θα πρέπει να έχει ένα ε, εσωτερικό μηχανισμό διακυβέρνησης, δημόσιο, έτσι ώστε να ε, εξασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις αυτές ε, θα βοηθούν στην επανισορρόπηση, στην εξορρόπηση μεταξύ των διαφόρων περιφερειών κάθε κράτους. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την φάση της επιλογής των έργων, θα συμφωνούσατε βασικό κριτήριο επιλογής να είναι η κοινωνική απόδοση που θα μετράτε με αντικειμενικό τρόπο από αντικειμενικούς εξωτερικούς εμπειρογνώμονες λαμβάνοντας υπόψη ε, το μοντέλο που επικρατεί, κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο που επικρατεί στις διάφορες περιοχές. I must apologize because I did not... Θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν κατάλαβα ακριβώ την πρώτη σας ερώτηση. and then... Θα απαντήσω πρώτα τη δεύτερη και αν επιτρέπει ο Πρόεδρος να ξαναεπαναλάβετε την πρώτη. Με χαρά θα την απαντήσω. Για τον ε, γενή εσωτερικό μηχανισμό, ναι. Θα φροντίσουμε να υπάρξουν δύο λεωφόροι προς αποφυγή του υπερβολικού κινδύνου σε μια χώρα. Είναι πάρα πολύ κοινό στη διαχείριση κινδύνου ε, η διασπορά των επενδύσεων και του χαρτοφυλακίου σε διάφορους τομείς και σε διάφορους κλάδους και γεωγραφικά. Ε, θα πρέπει λοιπόν οι επενδύσεις να μην γίνονται όλες ούτε στην ίδια χώρα, ούτε στην ίδια περιφέρεια, ούτε στον ίδιο κλάδο. Αλλά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους τομείς και κλάδους που έχουν ε, εντοπιστεί και επιλεγεί. Τώρα για τις ανισορροπίες. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων βασίζεται και εστιάζει στην προσθετικότητα. Το ξέρω ότι θα χρειαστεί να το επαναλάβω πολλές φορές και δεν θα κουραστώ γιατί είναι πραγματικά η κεντρική ιδέα και το κλειδί όλων αυτών που θέλουμε να κάνουμε, η προσθετικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στοχεύει σε έργα το Ταμείο στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, αλλά θα στοχεύει έργα που δεν μπορούν ήδη να ολοκληρωθούν αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τομέα. Αν υπάρχει ένα έργο το οποίο εκτελεί ιδιωτικός τομέας ή με οποιαδήποτε άλλη δημόσια επένδυση, δεν είναι επιλέξιμο κανονικά για το Ταμείο μας και έτσι στρέφεται προς κάποιες άλλες περιπτώσεις το Ταμείο και μπορεί, ελπίζουμε, να ε, καταργήσει τις ανεπισορροπίες. Και έχει να κάνει αυτό και με την κοινωνική ανάπτυξη. Και πάλι θέλω να φέρω εδώ το στοιχείο της προσθετικότητας και να σας πω τι προτείναμε. Το Ταμείο μας ακριβώς και πάλι στοχεύει σε έργα που φιλοδοξούν να προαγάγουν την κοινωνική ισορροπία. Με την άδεια του Πρόεδρου, θέλετε να επαναλάβετε την πρώτη σας ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση ήταν στην επιλογή των διαφορών έργων θα λυμφθούν υπόψη διάφορες, ε, διάφοροι όροι, διάφορες προϋποθέσεις και αν ένας από αυτούς θα είναι η, ε, η απαγόρευση, η δημόσια περιουσία δημόσια περιουσία, ε, περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου να χορηγείται ως ε, εγγύηση ή ενδεχομένως τα έσοδα τα οποία μπορούν να προκύψουν από δημόσιε δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα προσφερθούν στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων. Thank you. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θεωρούμε ότι μπορεί να προωθηθεί μόνο από τη στιγμή που κάποιος θα υποβάλει ένα συγκεκριμένο έργο. Αν χρησιμοποιούνται ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν δημόσια έσοδα, τότε αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή η κυβέρνηση, η διοίκηση σε μια χώρα έχει αποφασίσει μένα να κάνει κάτι τέτοιο. Από μόνο του σε καμία περίπτωση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν θα προωθήσει μία ατζέντα ιδιωτικοποίηση ε, Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Στόχο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων είναι έργα τα οποία προωθούνται είτε από τον ιδιωτικό είτε από το δημόσιο τομέα να υποβάλλονται ως έργα τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν, να χρηματοδοτηθούν από το ΕΦΣΥ. Πάντως εμείς δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο αυτό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά του ίδιου του δημοσίου, των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου. Μύρια Άντα, από την Επιτροπή Προπολογισμών, Οπόμε ομιλητής παρακαλώ. Ομιλήτρια. Μία-δύο ερωτήσει να κάνω και θα ήθελα και κάποιες διευκρινήσεις, ιδίως όσον αφορά την διάρθρωση του Ταμείου και τη σχέση που έχει το Ταμείο αυτό με τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα διαφορετικά ταμεία φοβάμαι ότι χρησιμοποιούνται ή ενδεχομένω να χρησιμοποιηθούν από ορισμένα κράτη-μέλη προκειμένου να προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτέ προκειμένου να έχουν στη συνέχεια πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ξέρετε ότι ορισμένα από τα διαφορετικά ταμεία έχουν ως στόχο να προωθήσουν το δημόσιο συμφέρον. Πολύ φοβάμαι όμως, είχα ανησυχούσα τουλάχιστον, αν κάποια κράτη-μέλη τα χρησιμοποιήσουν και να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις στα πλαίσια του EFSI. Τα κράτη-μέλη ενδεχομένως θα χρειαστεί να υποβάλουν χαμηλότερη συνεισφορά στο κοινοτικό προπολογισμό ακριβώς επειδή χρησιμοποιούν τα διευθυντικά ταμεία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να εκπονήσει κάποια νομοθετικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, ο οποίος ενδεχομένως να χρειαστεί να καταβάλει περισσότερα τέλη για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να του προσφέρονται, τουλάχιστον όπως το νερό ή η χρησιμοποίηση κάποιων αυτοκινητοδρόμων. Υπηρεσίες όμως που ανήκουν ήδη στο κράτος και παρέχονται από το κράτος ως δημόσιες υπηρεσίες. όσον αφορά το ζήτημα των ε, διαφορετικών ταμείων. Κοιτάξτε, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής και άμεσος. Πρόκειται για το τμήμα της ε, πρότασης, ε, για το οποίο εγώ λυπάμαι περισσότερο, διότι νομίζω ότι προκάλεσε πολύ μεγάλη σύγχυση, ενώ στην πράξη θέλαμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Στην πρότασή μας αναφερόμαστε σε μία διάταξη, η οποία αναφέρεται στη διασύνδεση μεταξύ διαρθρωτικών ταμείων και Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό το οποίο είναι σαφέ τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμεί θα θέλαμε μαζί σα να επεξεργαστούμε ενδεχομένω περισσότερο το κείμενο, τα διαρθρωτικά ταμεία πάντω δεν τροποποιούνται επουδενή μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ούτε ω προ τα κονδύλια του, ούτε ω προ τα κριτήρια επιλεξιμότητα τα οποία υπάρχουν για τα ταμεία αυτά τα διαφορετικά ταμεία εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αυτό είναι σαφέ, άρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε αυτό το πλαίσιο, μόνο για το δημόσιο δηλαδή συμφέρον. Εμεί σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι θα ανακατανείμουμε τι πιστώσει των διαφορετικών ταμείων προ κάτι άλλο το οποίο δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Τώρα στην πράξη. Αυτό το οποίο προβλέπουμε, όχι αποκλειστικά αλλά γενικά, είναι ότι υπάρχουν ορισμένα έργα τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν τη σήμερα ημέρα από, το, από τα διευθυντικά ταμεία, ενώ εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο λοιπόν βασίζεται όπως σας είπα στην προσθετικότητα. Αν μπορεί λοιπόν πλήρω να χρηματοδοτηθεί από τα μία, ταμεία, δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΕΦΣΥ. Αλλά μέσω του ΕΦΣΥ μπορεί να υπάρξουν άλλα έργα τα οποία θα καταφέρουν να χρηματοδοτηθούν ή να συγχρηματοδοτηθούν. Θα πρέπει πάντως τα έργα αυτά να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που υπάρχουν τόσο για τα δρατικά ταμεία, αλλά και τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία θα ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, δηλαδή το κριτήριο προστατικότητας και ενδεχομένω και άλλα κριτήρια. Τώρα, πώς προστατεύουμε το φορολογούμενο σε σχέση με έργα τα οποία τον αφορούν άμεσα. Ξέρω ότι πολλές φορές ε, με 28 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα διαφέρουν πολύ. Για ορισμένα κράτη-μέλη, ορισμένες υπηρεσίες ή έργα αφορούν άμεσα τον φορολογούμενο και παρέχονται από το κράτος, άλλες πάλι χώρες τα πράγματα είναι διαφορετικά και υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός ιδιωτικοποίησης. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κανένα έργο δεν μπορεί να υποβληθεί αν δεν έχει την υποστήριξη των ίδιων των ανάδοχων του έργου αυτού. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς από μόνοι μας και ως χειριστές του ΕΦΣΥ να σπρώξουμε ένα έργο από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Η Ελέσια Μόσκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να αναφερθώ σε ένα σημείο το οποίο αναφέρθηκε πολλές φορές αλλά για το οποίο τελικά βλέπουμε ότι δεν δόθηκε συγκεκριμένη απάντηση και πολλοί ανησυχούν. Ελοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν περισσότερες ανισότητες ανάμεσα σε χώρες οι οποίες έχουν οικονομική άνεση και χώρες οι οποίες υποφέρουν οικονομικά. Να διατυπώσω λοιπόν ένα ερώτημα το οποίο είχα υποβάλει γραπτός. Θα θέλα να είχα περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το ερώτημα αυτό. Σας ρωτούσα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να διευρυθεί το πεδίο εφαρμογή της ρήτρα ε, επενδύσεων όσον αφορά το τμήμα εκείνο που αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μας δώσατε αρνητική απάντηση. Εφόσον λοιπόν δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο και να χρησιμοποιήσουμε τη ρήτρα αυτή την επενδυτική, πιστεύετε ότι υπάρχουν ε, άλλοι μηχανισμοί που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την πρώτη ερώτηση, τον κίνδυνων διαφορών. Καταρχήν έχουμε το θέμα της ε, προσθετικότητας, δεν θα τα επαναλάβω. Ένα άλλο όμως στοιχείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην πρόταση της Κομισιόν, είναι το κέντρο επενδύσεων. Το επενδυτικό κέντρο. Στην πρότασή μας εργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να προτείνουμε την δημιουργία μιας ενιαίας θηρίδας για τεχνική συνδρομή στην Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε ότι οι χρηματαγορές στην Ευρώπη εξελίσσονται διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Και η χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων απαιτεί εξειδικευμένη βοήθεια. Για αυτό το λόγο θα έχουμε αυτή την ενιαία θηρίδα για να προσφέρει την κατάλληλη τεχνική συνδρομή που, χρειάζεται, ε, που χρειάζονται όσοι προτείνουν υποβάλλουν κάποιο έργο. Δεν, μας, δεν θέλουμε να αυξηθούν οι διαφορές τα κενά. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι διαφορές ανάμεσα σε χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του συστήματος προτιμήσεων, και την προτιμησιακή μεταχείριση. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι σημαντικό για πολλούς από εσά. Δεν προτείναμε την αλλαγή του κανονισμού. Προτείναμε απλώς να τον, να τον ερμηνεύσουμε όσο πιο φιλικά γίνεται. Βέβαια, υπάρχουν και όρια σε αυτό, διότι θα πρέπει να τηρηθεί το κείμενο η ουσία του κειμένου. Είμαστε πεπισμένοι ότι η μεταχείριση την οποία προτείνουμε θα επιτρέπει τις υγιείς επενδύσεις συνδυαζόμενα συνδυαζόμενες με τη δουλειά το, της επενδυτικής πλατφόρμας. Αν τα κράτη-μέλη θέλουν να αυξήσουν το επίπεδο των επενδύσεών τους, θα, το σύστημα θα το επιτρέψει. Χωρίς να χρειαστεί να παραβούμε τους κανόνες που έχουμε για την γεωγραφική κατανομή και χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε τον κανονισμό του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Ευχαριστώ κύριος Λούκε. Καταρχάς, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στη συνέχεια οι εγγυήσει είναι ενισχύσεις και δεν ισχύει εδώ το άρθρο 107 της Συνθήκης για την απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων και στο βαθμό που ε, παραπέμπεται στις εξαιρέσεις ε, μιλάμε για 315 δισεκατομμύρια επενδύσεων ε, που είναι προς όφελος ε, του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Αυτό εμένα μου φαίνεται αφισβητήσιμο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε σχέση με την ενίσχυση αυτών θα ήθελα να ρωτήσω πώς αυτή συνδέεται και συσχετίζεται με την ουδετερότητα στον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Στο άρθρο 125 αναφέρεστε, όχι, στο 107. 107 άρθρο της συνθήκης. Α, 107, μάλιστα. Thank you. Ευχαριστώ. Κρατικές ενισχύσεις. Προφανώς είναι ζήτημα κομβικό και αυτό που πρέπει να δούμε. Είμαι βεβαίως ότι διαβάσατε στην πρόταση την αιτιολογική σκέψη που αναφέρεται στην ανάγκη να είμαστε συνεκτικοί με τα όσα ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις. Θα πρέπει να βρεθεί μια λεπτή ισορροπία. Από τη μια θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα κρατικά χρήματα από τις συνεισφορές του κοινοτικού προϋπολογισμού δεν σπαταλώνται, δεν διασπαθίζονται και δεν υπερ, σπαταλώνται ή μάλλον καταναλώνονται για έργα αλλά δεν θα πρέπει να εξαιρούνται και πάρα πολλά έργα από τον έλεγχο κρατικών ενισχύσεων. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφής. Θέλουμε να παραμείνουμε σύμφωνοι με τα όσα ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις και αν μου επιτρέψετε πώς το βλέπουμε στην πράξη, να επεκταθώ λίγο παραπάνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει, θα εκδώσει μια ανακοίνωση σχετική με τις κρατικές ενισχύσεις και πώς αυτές εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα υπάρχουν αρχές υψηλό επίπεδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται τα χρήματα ε, που θα δαπανώνται με την υποστήριξη του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Δηλαδή όχι υπερβολική αποζημίωση, όχι επικάλυψη υφισταμένων έργων και άλλα τέτοια έργα, κριτήρια. Σε πολύ περιορισμένο όγκο από πλευράς ποσών. Και θα θέλαμε να γίνονται πάντα σεβαστά αυτά. Δηλαδή δεν μπορείς να χτίσεις ένα αεροδρόμιο 10 μέτρα από το διπλανό, από το προηγούμενο, ούτε ε, αυτό εξυπηρετεί τους στόχους της βιωσιμότητας και στην ανάπτυξη ε, του στόχου του Ταμείου εννοώ. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό. Η εθνική συγχρηματοδότηση και η στήριξη όλοι γνωρίζετε, ανάγεται ε, και μάλλον ελέγχεται με μια απλή δοκιμή για τις κρατικές ενισχύσεις και χρειάζεται και πολύ χρόνος, ένα έτος συνήθως. Και γιατί θα πρέπει να γίνεται στην κορυφή αυτός ο έλεγχος στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Έτσι ώστε οποιαδήποτε παράλληλη ε, ε, επένδυση ή χρηματοδότηση να γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Και το μόνο που θα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, η απουσία υπερ ε, αποζημίωσης. Δηλαδή, από το τον εκτενή έλεγχο και το ενδελεχεί που χρειάζεται ένα χρόνο, τελικά θα χρειάζονται λίγες εβδομάδες. Και πολύ πιο γρήγορα θα προχωρεί το έργο, ε, που δεν θα προχωρούσε αν γινόταν πλήρης ε, συστηματικός έλεγχος για τις κρατικές ενισχύσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση για τα μέσα και το Ταμείο Εγγύησεων. Ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι για το Ταμείο Εγγύησεων δεν ε, θεωρούν ε, ε χρήσιμο να συνδεθεί με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς, ε, γιατί ούτε τα διορθωτικά ταμεία ούτε τα άλλα μπορούν να συνδεθούν με αυτό. Ε, και το πήραν από το Horizon και από την Connect Europe. Το είπε και ο συνάδελφος Έλερ, είναι 1 προς 13 ο πολλαπλασιαστής για ε, προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Εδώ έχουμε ένα μοχλό 1 προς 15 και άκουσα σήμερα ότι είναι λέει και μέσος όρος, ότι μπορεί να είναι και λιγότερο από 15. Μα αν κοιτάξουμε τα έργα, νομίζω συχνότερα θα είναι λιγότερο από 15, παρά 15. Μήπως Ε, ε, και μήπως ε, δεν είναι πάρα πολύ φρόνιμο να θυσιάζουμε έναν ασφαλή τρόπο υπολογισμού και μοχλό 1 προς 13 στο βωμό του 1 προς 15 που δεν είναι τόσο ασφαλής. Επίσης τα έργα αυτά που μας απασχολούν έχουν υψηλό κίνδυνο γι' αυτό το λόγο υπάρχει και το Ταμείο Εγγυήσεων. Παρ' όλα αυτά οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να φέρουν τουλάχιστον ένα πολλαπλασιαστεί της τάξης του 5. Ε, αλλά για να το κάνουν αυτό οι ιδιώτες πρέπει να έχουν και ένα ορατό κέρδος. Ε, υπάρχει ένα κλάστερ απόδοσης, δηλαδή τι απόδοση θα έχει επέβησή του κάθε ιδιώτη. Έχει υπολογιστεί αυτό. Και θέλω να πω και αναφερόμενοι στον εισηγητή. Όταν πρέπει να εκτελούνται μεγάλα έργα, ας πούμε ένα έργο υποδομής μεταφορών, στα κράτη-μέλη χρειάζονται μακροχρόνιες διαδικασίες έγκρισης. Τι θα γίνει και αυτό θα το περάσετε σε fast track, το έχετε προβλέψει αυτό για την ταχεία διεκπαιρέωση. Και τι γίνεται με τους εθνικούς φορείς. Εγώ ε, ήμουν ε, επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβολίο, στο εποπτικό μάλλον της ε, Αυστριακής Αρχής για την Ανάπτυξη ε, και Αυτές οι αναπτυξιακές αρχές, οι δομές μπορούν να συντονίζουν, να ελέγχουν, αλλά πώς θα συνεργάζονται με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτά τα έχετε προβλέψει, έχετε προτείνει αντίστοιχες διατάξεις. Commission. Η Επιτροπή. Καταρχήν, πράγματι, κάτι σημαντικό για τον πολλαπλασιαστή 15 δεν είναι κάποιο αβέβαιο πολλαπλασιαστή. Εγώ ε, ηθελημένα είπα ότι ε, δεν ε, θα εξασφαλίζει το 15 κάθε έργο. Αλλά όχι επειδή ε, δεν θα είναι βέβαιο. ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος και βέβαιος. Τον έχουμε θέση και, θα τον... και είμαστε πεπισμένοι ότι θα καλυφθεί μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μερικέ φορέ θα είναι υψηλότερο, μερικέ φορέ ε, χαμηλότερο. Αλλά αυτό οφείλεται στη φύση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν. Το ΕΦΣΥ, το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, θα έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα έργων. Ορισμένα από αυτά οδηγούν με φυσικό τρόπο σε υψηλό πολλαπλασιαστή, αλλά σε χαμηλότερο πολλαπλασιαστή. Γι' αυτό το λόγο και είναι σκόπιμο αυτό το εύρος ε, ε, έργων δεν αναζητούμε τον ίδιο πολλαπλασιαστή για όλα τα έργα αλλά ένα μέσο όρο τον οποίο τον έχουμε καθορίσει το 15% για να πετύχουμε το στόχο των 315 δισεκατομμυρίων. Τώρα, ψηλό κίνδυνος και τι έχει να κερδίσει ο ιδιωτικός τομέας. Ναι, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων στοχεύει στα πιο επισφαλή έργα, αλλά σίγουρα θα είναι βιώσιμα από οικονομικής πλευράς έργα. Δεν θα χρηματοδοτούνται έργα τα οποία δεν δείχνουν να είναι βιώσιμα. Και η Επενδυτική Επιτροπή θα διασφαλίσει αυτό ακριβώ το κριτήριο. Μόνο έτσι θα μπει μερικά του χρηματοδιωτικό τομέα. Τώρα, ο ιδιωτικό τομέας δεν είναι καλοί σαμαριτές, περιμένουν κέρδη. Αυτά όμως είναι έργα ναι, που θα θέλαμε να χρηματοδοτήσει έτσι και αλλιώ ο ιδιωτικό τομέα από μόνος του, αλλά δεν είναι διατεθειμένος πρόθυμο να τα χρηματοδοτήσει μακροπρόθεσμα. Αποφεύγοντα το επικίνδυνο τμήμα είναι προφανές ότι ε, απαρνούνται και τα υψηλά, την υψηλή κερδοφορία. Ε, δεν θα έχουν τόσο υψηλή κερδοφορία αυτά τα έργα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συντονισμό με, άλλα, με άλλους μηχανισμούς. Έχουμε δύο επίπεδα για να το εξασφαλίσουμε. Ένα εκ των προτέρων, ένα εκ των υστέρων. Ο εκ των προτέρων προληπτικός συντονισμός θα γίνεται μέσω της Επενδυτικής Επιτροπής. Έτσι κι αλλιώς θα γίνονται οι έλεγχοι που γίνονται πάντοτε, αλλά επιπλέον όταν κάποιος προτείνει, υποβάλλει ένα έργο και λέει δεν μπορώ να το χρηματοδοτήσω, μόνος μου αναζητώ χρηματοδότηση από αλλού, θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση από αλλού. Αν η Επενδυτική Επιτροπή θεωρήσει ότι υπάρχει άλλος μηχανισμός, άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο για να το χρηματοδοτήσει, δεν θα δεχτεί αυτό το έργο. Τώρα για τον εκ των υστέρων ε, έλεγχο. Στην, ε, στο άρθρο 10 για τις εκθέσεις. Ίσως δεν, δεν δώσαμε αρκετή ε, σημασία στο 10.2α που είναι ε, αναπόσπαστο τμήμα της πρότασής μας. Αφορά την αξιολόγηση του πού δαπανήθηκαν τα κονδύλια και πώς. Και αυτό, αυτός, αυτή η αξιολόγηση θα αφορά όλα τα κοινά έργα, όλα τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό. Έτσι ώστε ε, να μην υποκαθιστά το ένα το άλλο και να ε, μπορούν να έχουμε αλληλοβοήθεια. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες ερωτήσεις έχω και εγώ που έχουν να κάνουν περισσότερο με θέματα πολιτικής και κάποιες ερωτήσεις μου είναι και τεχνικής φύσης. Νομίζω ότι η λίστα ήταν να είχαμε πιο ανταγωνιστικές οικονομίες, έτσι θα λύναμε και το οικονομικό μας πρόβλημα. Αυτό όμως σημαίνει ότι κάποια κράτη πρέπει να κάνουν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Πρώτον ερώτημα λοιπόν. Από τεχνική πλευρά θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων με την υποχρέωση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για ορισμένε χώρε. και κατά αυτόν τον τρόπο να σεβαστούμε όμω και τι αρμοδιότητε των κρατών μελών. Δεύτερον, στον κανονισμό προβλέπεται ότι το ΕΦΣΥ θα έχει μόνιμο καθεστώς. Για ποιο λόγο? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χρησιμοποιήσει το ταμείο αυτό προκειμένου να ξεκινήσει μια περαιτέρω συζήτηση όσον αφορά για παράδειγμα του Ιδίου, πόρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Τρίτον, στο άρθρο 8 λέγεται ότι τα πλεονάσματα θα πάνε στο γενικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερώτημα προς αυτό. Γιατί δεν θα ήταν πιο λογικό να πάνε τα πλεονάσματα αυτά στα ίδια τα ταμεία. Μια ερώτηση πρακτικής φύσης όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Κέντρο Επενδύσεων εν μέρη θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα. Μήπως είναι κάπως υψηλό αυτό το ποσό. Μία ακόμη ερώτηση. Μήπως, διακόπτει ο Πρόεδρος, πολλές ήταν οι ερωτήσεις σας. Μήπως να δοθούν πρώτα κάποιες απαντήσεις. Μα η τελευταία μου ερώτηση ήταν κύριε Πρόεδρε. Για ποιο λόγο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θέτει ένα κατόφλι επιχειρήσεων που έχουν 3.000 εργαζομένους. Πώς επιλέξατε αυτό το κατόφλι 3.000 εργαζόμενοι. Πέντε πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω γρήγορα. Αν θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να συνδεθεί με τις δραστηριοτικές μεταρρυθμίσεις. Οι δραστηριοτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση σίγουρα, το λέμε αυτό και στην έκθεση. Αν όμως συνδέσουμε την υποστήριξη από το Ταμείο αυτό με τις γραφικές μεταρρυθμίσεις, τότε προκύπτει και ένα επόμενο στοιχείο, ο χρόνος και το κόστος. Τόσο σε εθνικό επίπεδο, αλλά όσο και στον τρίτο πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου, θα μπορούσε να γίνει η διασύνδεση αυτή. Παρ' όλα αυτά δεν θα την κάνουμε ακριβώ επειδή μιλάμε για διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και διαφορετικά ποσά. Όσον αφορά την μόνιμη φύση το μόνιμο αυτό καθεστώ του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και ο τύπο έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα αυτό. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που προτείνει είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να διονυστεί μόνο αν στεφθεί με επιτυχία. Μόνο 60 δισεκατομμύρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αν όμω χρησιμοποιηθούν, θα μπορούσαν τουλάχιστον να συμπληρωθούν με την απόδοση των επενδύσεων, με επιπλέον κέρδη που θα πράττουν στο μέλλον. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι, οκ, ας α, είναι μόνιμη φύση του εύση αρκεί να παράγει κέρδη. Αν για οποιοδήποτε λόγο αποτύχει το εύση, τότε προφανώς δεν θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Επομένως, κατά αυτόν τον τρόπο δίνεται ένα κίνητρο σε όλους τους συνεισφέροντες να εγγυθούν την επιτυχία του ΕΦΣΥ. Τώρα αν τα πλεονάσματα θα πρέπει να πηγαίνουν στο γενικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί προβλέπετε αυτό. Κοιτάξτε, αναφέρεστε σε μία διάταξη η οποία αρχίζει και ισχύει μόνο αφού ξεκινήσουν οι αναθεωρήσεις των προγραμμάτων. Είχαμε σκεφτεί ε, τη χρησιμοποίηση των κερδών με διαφορετικό τρόπο στον κοινοτικό προπολογισμό. Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποσαφηνίσουμε το εξή. Μιλάμε, για Μιλάμε για μακροπρόθεσμε βιώσιμε επενδύσει στην Ευρώπη. Δεν λέμε αυτή τη στιγμή θέλουμε να κάνουμε κέρδη τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αναφερόμαστε σε συνεχή κερδοφορία για τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώ το λόγο θεωρούμε ότι θα έχουμε πάρα πολλέ ευκαιρίε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να κάνουμε προσαρμογές σε διάφορες διατάξεις αφού μάλιστα ολοκληρωθούν και οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτά τα 20 εκατομμύρια για μας δεν αποτελούν στόχο. Εμείς είπαμε έως 20. Αυτό έχουμε συμφωνήσει και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για μας δεν είναι υπερβολικό το ποσό αυτό, ακριβώς επειδή δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Μέσω του ταμείου αυτού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεφιστάμενα τεχνικά μέσα, αλλά και την επιπλέον τεχνική υποστήριξη που μπορεί να υπάρχει, τόσο για το ΕΦΣΥ, όσο και για να παραχθεί όχι μόνο τεχνική υποστήριξη στο Λουξεμβούργο, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και τεχνική υποστήριξη εκεί που απαιτείται περισσότερο, δηλαδή στο επίπεδο της, ε, του ίδιου του έργου, εκεί πέρα δηλαδή που υλοποιείται το έργο. και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε νομίζω να περιφυροποιήσουμε περισσότερο την συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνεχίσει να βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, αλλά νομίζω ότι πολλοί συμμετέχοντες τώρα, πολλοί ενδιαφερόμενοι, μπορούν να έχουν πιο άμεση πρόσβαση και σε περιφερειακό επίπεδο. Όσον αφορά το όριο αυτό των 3.000 εργαζομένων. Κοιτάξτε, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στην κοινοτική νομοθεσία, ένα τέτοιο κατόφλι σε άλλα σημεία, σε άλλες κοινοτικές νομοθεσίες. Δεν υπάρχει ανώτατα αυτή οροφή. Πάντως έχουμε 75 δισεκατομμύρια ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν όμως υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν εργαζομένους άνω των 3.000 τότε μπορούν να απευθυνθούν στο τμήμα καινοτομία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και να χρηματοδοτηθούν από εκεί. Δεν προσπαθούμε λοιπόν να αποκλείσουμε κάποιες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ο κ. Φερνάνδη από την Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τον άλλο εισηγητή, τον συνάδελφό μου, και να ευχαριστήσω την Κομισιόν ε, που είναι πραγματικά άξια ε, και δέχτηκε να συμμετάσχει σε αυτό το μαραθώνιο ερωταποκρίσεων. Και ε, είναι πολύ ωφέλιμες αυτές οι απαντήσεις. Το ταμείο αυτό θα είναι πρόκληση και για τους επενδυτές αλλά και για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Άλλωστε πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ποσό, 315 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μην ξεχνάμε τη στήριξη που θα δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ε, διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς με την άρση των εμποδίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξή. Τι επίπτωση περιμένετε ότι θα έχει στη δημιουργία θέσεων απασχόληση, στην αύξηση του ΑΕΠ και στην ανάπτυξη το ταμείο αυτό. Ε, τι επίπτωση θα έχει στην άρση των φραγμών και στην εμβάση της εσωτερικής αγοράς και τρίτον, τι επιπτώσει θα έχει το Ταμείο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαιτέρως στις επιχειρήσεις ε, έρευνας και καινοτομίας. Ευχαριστώ. Commission. Ευχαριστώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. Impact. Σε ό,τι αφορά τι επιπτώσεις των, του επενδυτικού σχεδίου γενικότερα, Ε, ήταν η πρώτη από τις 110 που μας ε, στείλατε. Δημιουργία 1 ως 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αύξηση του ΑΕΠ ε, κατά 340-410. Από 330 410, συγγνώμη. Να σας εξηγήσω. η Κομισιόν χρησιμοποίησε το μοντέλο τη με τις υποθέσει εργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, πρόκειται για ένα μοντέλο ε, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν ε, υπό την προπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί πλήρης προσθετικότητα. Γι' αυτό το λόγο την υπογραμμίζουμε την προσθετικότητα. Σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ένα από τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου είναι να δοθεί βοήθεια ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό το λόγο προτείναμε τη δημιουργία αυτού του παραθύρου στόχου 75 δισεκατομμυρίων με στόχο της μικρομεσαίας επιχειρήσεις και της επιχειρήσης μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ε, Είμαστε στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για του υπολογισμού αυτούς. Αλλά από αυτά τα 75 δισεκατομμύρια θέλουμε να δώσουμε χρηματοδότηση σε 80.000 περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Με πρόθεση, χάρη στη σημασία τους ε, στην οικονομία, να ε, δώσουμε μια ιδιαίτερη όθηση στι καινοτόμε επιχειρήσεις. Αυτά τα νούμερα έχουν ληφθεί υπόψη στο, στο συνολικό υπολογισμό ε, για τις θέσεις εργασίας και την αύξηση του ΑΕΠ. Σας ευχαριστώ. Πριν ολοκληρώσουμε, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το γύρο ερώτα απαντήσεων που ήταν πάρα πολύ εντατικός. Φυσικά δεν διαπραγματευόμαστε εμείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας, κάνει απαντήσεις, μας δίνει απαντήσει συγγνώμη για την πρότασή τους. Στη συνέχεια η ε, πρότασή τους θα συζητηθεί αλλού και θα δούμε τι ε, θα αποφανθούν οι συνομοθέτες. Πάντως είναι πολύ καλό να έχουμε διευκρινήσει σε αυτή την τεχνική συνεδρίαση για την πρόταση, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία ε, όπου είναι θεμητές και κάποιες αμφιβολίες μας. Γι' αυτό θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Σωστά απαντήσατε στην ε, απάντηση 84 ότι οι εγγυήσει θα δίνονται υπό όρου που θα έχουν αποφασίσει οι σύνομοθέτε. Ναι, ωραία. Αλλά αυτό γνωρίζουμε ότι δεν γίνεται με άμεσο τρόπο, δεν είναι δυνατό. Για μια σειρά από περίπλοκους λόγους, το καταλαβαίνω ότι δεν έχει και νομική προσωπικότητα το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το καταλαβαίνω, αλλά δεν αυξάνεται και το κεφάλαιο ε, προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οπότε χρειάζεται μια διαφορετική δομή. Με αυτόν τον κανονισμό λοιπόν τι δημιουργούμε. Ένα γενικό πλαίσιο για μια συμφωνία που θα πρέπει να ε, επιτευχθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και μέχρι τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος θα είναι αυτός ο κανονισμός βάσει της κείμενης πρότασης και ποιο θα είναι το δικαίωμα των συνομοθετών να το καθορίζουν όλα αυτά. Και όπως λέτε και στην απάντησή σας υπαριθμών 30, η Επενδυτική Επιτροπή θα ακολουθεί συγκεκριμένες ε, κατευθυντήριες γραμμές που θα τις δίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ε, αυτό δεν είναι ακριβώς ε, αρμοδιότητα των συνομοθετών. Δηλαδή δεν θα έχει λόγο η δημοσιονομική αρχή και αυτό μπορεί να αποτελεί πρόβλημα. Εσείς το βλέπετε τουλάχιστον ως πρόβλημα. Το έχετε εντοπίσει. Και ένα δεύτερο έχει να κάνει με την εγγύηση. Ο όρος να δοθεί εγγύηση είναι η βιωσιμότητα του έργου. Είναι πάρα πολύ ισχυρή αυτή η διατύπωση. Είστε όμως βέβαιοι ότι η βιωσιμότητα ενός ε, έργου που εκτιμάται από μια Επιτροπή Επενδύσεων που οι ειδικοί ε, έχουν ειδίκευση αποκλειστικά στη χρηματοδότηση έργων γιατί θελήσατε να είναι πάρα πολύ στενό το πεδίο αρμοδιοτήτων. Πώς θα το καταφέρει αυτό και ότι είναι προσθετική και συνάδει με το γενικότερο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να μειωθούν οι διαφορές, να υπάρξει ε, αποτελεσματική συνεισφορά στους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Αυτό είναι αποκλειστικά στα χέρια μιας χούφτας ανθρώπων που έχουν εξειδίκευση στη χρηματοδότηση έργων. Πώς θα τα κρίνουν όλα αυτά και πώς θα τα αξιολογήσουν. Αυτό δεν σας φαίνεται πρόβλημα. Ε, και πώς εκεί θα δράσει και θα αποφανθεί ο συνομοθέτης. Yes. Μάλιστα. Ενδεχομένως να μακρηγορήσω λίγο στην απάντησή μου για το πρώτο σας ερώτημα. Έχουμε προφανώς τα τρία επίπεδα, τον κανονισμό, τη συμφωνία την οποία πρέπει να συνάψουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων και έχουμε και τις πολιτικές στη συνέχεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρώτον, πρέπει να ακολουθήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Σε καμία περίπτωση η συμφωνία Εύση δεν μπορεί να αντιβαίνει στον κανονισμό. Και οι πολιτικές του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν προφανώς να αντιτάσσονται είτε στη συμφωνία είτε στον κανονισμό. Πρέπει να πετύχουμε δηλαδή την κατάλληλη ισορροπία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της πρότασής της πρότεινε ένα σενάριο ισορροπίας αν θέλετε και οι συνομοθέτες για διάφορους λόγους είπαν ότι η ισορροπία αυτή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι η κατάλληλη για αυτούς και ενδεχομένως να θέλουν να προσθέσουν κάποια επιπλέον στοιχεία στα πλαίσια της συμφωνίας ή στα πλαίσια του κανονισμού. Εμείς βέβαια προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία μαζί σας, προκειμένου να συμπεριλάβουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλετε να δείτε στον κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όντως τα έργα τα οποία θα επιλέξουμε συνάδουν και με τις δικές σας, τις, α, τους δικούς σας τους στόχους, τα δικά σας τα μελήματα. Τώρα, όσον αφορά την Επιτροπή Επενδύσεων και αν η εμπειρογνωμοσύνη που έχουν σε θέματα χρηματοδότηση επενδύσεων αρκεί για να αξιολογήσουν σωστά τα προτινόμενα έργα. Κοιτάξτε, είχατε τη δυνατότητα να δείτε το προσχέδιο της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στην οποία λέμε ότι ε, η Επιτροπή Επενδύσεων θα θέλαμε να έχει τα εξή δύο βασικά χαρακτηριστικά και μια ευρή εμπειρία σε αυτά. Πρώτον, γνώσεις για διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες στην Ευρώπη. Θα πρέπει τα μέλη δηλαδή, της Επιτροπής αυτής όντως να έχουν συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη για διάφορες περιοχές της Ευρώπης, αλλά και δεύτερον για διάφορους τομείς. Αν και πάλι τώρα οι συνομοθέτες θέλουν να περάσει το κριτήριο αυτό στον κανονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας προκειμένου να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας αυτήν και για όλες τις προηγούμενες απαντήσεις. Νομίζω ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτησή μας και να και τώρα στους συνομοθέτες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εργαστούν και να παρουσιάσουν το πρώτο επίσημο σχέδιο πρότασης. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύε τη συνεδρίαση.